Colleagues, uh, if you could take your seats, please. Thank you. Καλημέρα, συνάδελφοι. Ξεκινάμε με την αποδοχή της ημερήσιας διάταξης. Το 15 για την προφορική ερώτηση του Ντεπρέ Η συζήτηση θα γίνει ε, μετά το 21. Αν δεν υπάρχουν ε, ε, αντιρρήσεις, τροποποιείται η μερίσια διάταξη. Για το σημείο 2 τώρα, πρακτικά της 19ης Οκτωβρίου, 30 Σεπτεμβρίου και αυτά θεωρούνται δεκτά, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Σημείο 3. Για τις γλώσσες δυστυχώς κελτικά δεν έχουμε. Και μετά έρχομαι τώρα στις συστάσεις των συντονιστών για τον ορισμό εισηγητών, Σκά Κέλλερ των Πρασίνων, εισηγήτρια για την απόφαση του Συμβουλίου 2.20 για τη διεθνή προστασία. Ο κύριος Μέρα θα είναι επίσης ε, υπεύθυνο για το πακέτο το διπλό ευφυ, σύνορα. Λοιπόν, αυτές είναι οι συστάσεις των συντονιστών. Το τρίτο σημείο, συνάδελφοι, είναι η Επιτροπή ΣΕΝΤΙ και εμείς σήμερα το απόγευμα στις 3 έχουμε στο PHS 5.001 ακρόαση για την διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης καταπολέμηση της ε, εμπορίας ανθρώπων. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε την ακρόαση αυτή. Ξέρω βέβαια ότι όλοι έχετε πάρα πολλή δουλειά αλλά θα ήταν καλό να μπορέσουμε να είμαστε παρόνες και θα σας ήμουν ευγνώμων αν πράγματι είμαστε παρόντες. Γιατί υπάρχουν πολλά θέματα γύρω από αυτό που μας ενδιαφέρουν. Η παρουσία μας θα εκτιμηθεί δεόντως. Και τέλος, άλλο ένα συνοπτικό αλλά σημαντικό θέμα. Είδατε ότι τα έγγραφα της Επιτροπής δεν είναι διαθέσιμα πλέον. Αυτό αποφασίστηκε από τους συντονιστές μαζί με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Δεν έχουμε συστηματική διανομή των εγγράφων πλέον, αλλά μπορείτε να τα ζητήσετε αν θέλετε από τους κλητήρες. Αυτό το κάνουμε για να μειώσουμε τα χαρτιά που χρησιμοποιούμε. Να μειώσουμε το κόστος και να είμαστε φιλικοί περιβαλλοντικά. Αν κάτι σας λείπει λοιπόν ζητήστε το. Αν έχετε ανάγκη από κάτι σε έγγραφο μπορείτε να το ζητήσετε από τους κλητήρες. Περνάμε στο σημείο 4 για την εκπαίδευση των δυνάμεων στον τομέα τον δικαστικό. Ο κύριος Δίας Ντεμέρα μπορεί να κάνει μία μικρή εισαγωγή σε λίγο, αλλά πρόκειται για μία φάση δεύτερης ανάγνωσης. Ενθυμίστε ότι στην πρώτη ανάγνωση, την προηγούμενη εβδομάδα, έγιναν ανεπίσημες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. November. So we now start the Ξεκινάει τώρα η επίσημη διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Διάς θα μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν μακρότατες διαπραγματεύσεις. Οι κανόνες είναι ξεκάθαρες. Είναι ξεκάθαροι λοιπόν οι κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα και αυτό θα το διευκρινίσει και ο εισηγητής σε λίγο. Η προθεσμία είναι 21η Απριλίου και η ψηφοφορία θα γίνει στις 28 Απριλίου. Θα δώσω το λόγο πλέον στον εισηγητή μας, Έχετε το λόγο κύριε Διαστεμέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ των προτέρων θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί σωματικά δεν είμαι και πάρα πολύ καλά. Αλλά θα κάνω μία προσπάθεια για να κάνω την ανακοίνωση που οφείλω. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και τρία χρόνια προσπαθούμε να προχωρήσουμε στον σημαντικό αυτό κανονισμό και στα πλαίσια του τριγωνικού διαλόγου καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική ε, λύση το Νοέμβριο ε, του 2015. Θα ήθελα λοιπόν να προχωρήσουμε στην δημιουργία νομικά ενός οργάνου υψηλής χρησιμότητας ε, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως η υπηρεσία που ασχολείται με τον έλεγχο του ίντερνετ κτλ. Έχουμε ενισχύσει τις αρμοδιότητες της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στο πρώτο παράρτημα της έκθεσής μας. Ταυτόχρονα και εκ των υστέρων μάλλον η θέση του Συμβουλίου είναι αυτή που συμφωνήσαμε τον Νοέμβριο, έγινε επίσημα δεκτή στις 3 Μαρτίου του 2016 και απεστάλλει εκ νέου στο Κοινοβούλιο όπως το είπε και ο Πρόεδρος πριν. Η θέση αυτή, την οποία μπορώ να χαρακτηρίσω κοινή θέση και με την οποία σύμφωνο, μπορεί να τροπολογηθεί από την Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ μέχρι τις 21 Απριλίου και θα πρέπει να ψεφιστεί από πλευράς μας την εβδομάδα ε, την επόμενη, 28 Απριλίου. Θα μπορούσε λέω, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάντως μπροστά μας μια συμφωνία η οποία είναι σταθμισμένη, έχει συζητηθεί επί μακρόν και πράγματι είναι πολύ συνενετική και αυτό έγινε ε, χάρη ακριβώς στην τεράστια προσπάθεια που έκαναν όλες οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν και τις απόψεις των συναδέλφων και των σκιωδών. Θέλω να τους ευχαριστήσω και να τους μεταφέρω τα αισθήματα ευγνωμοσύνης που τρέφω απέναντί τους και σας ζητώ στις 28 Απριλίου να υπερψηφίσετε το κείμενο αυτό έτσι ώστε να φτάσουμε στην Ολομέλεια τον μήνα Μάιο. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη και αυτό ακριβώς το λόγο το μέσο αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής. Εν κατακλείδη θα ήθελα να μου ξαναδώσετε ίσως τον λόγο αφού ομιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι που το επιθυμούν. Absolutely, I'll, I'll give... Θα σας δώσω το λόγο στο τέλος να ολοκληρώσετε κυρία Διαστεμέρα. Πάμε στους Κιώδης. Τζο Βάιντεν για τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τον εισηγητή. Πιστεύω πως είχαμε μια πολύ καλή και επικοδομητική συνεργασία τα τελευταία τρία χρόνια που ε, βασίστηκε στην παρακολούθηση των εξελίξεων. Ε, χαίρομαι που καταφέραμε να αντιδράσουμε σχετικά γρήγορα στις εξελίξεις και δείξαμε την ανάγκη ευελιξία έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Ε, σίγουρα Υπήρξαν κάποια προβλήματα, όμως ε, αυτά θα επιληθούν, πιστεύω, νομοθετικά, έτσι ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους αυτήν την πάρα πολύ καλή νομική βάση που έχουμε κερδίσει με την αξία μας. Thank Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ναι. Τίμωθη, έχεις το λόγο. Τίμωθη Θα ήθελα και εγώ να στηρίξω τον εισηγητή και τη δουλειά που έχει κάνει. Ιδιαίτερα αφού ε, εκτιμούμε όλη τη δουλειά της Ευρωπόλ, δεδομένων των απειλών που έχουν παρουσιαστεί, πιστεύω ότι μας επιτρέπει το παρόν μέτρο να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία. Επίσης πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ στην προστασία των δεδομένων και στα δικαιώματα του ατόμου, του πολίτη στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο μας απασχολεί και μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, έχω εμπειρία σε αυτό το θέμα. Είναι κάτι που συζητούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και πιστεύω πως πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση και να στηρίζουμε το έργο της Ευρωπόλ. Γι' αυτό λοιπόν θα δείξω τη στήριξή μου στον εισηγητή και ελπίζω να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Ο σχεδόν εισηγητής από την Άλντα, κύριος Πίτερσον. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία με όλες τις πολιτικές ομάδες και διότι περασπίστηκε τη θέση του Κοινοβουλίου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δείχνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη ε, και πιο ολοκληρωμένη αστυνομική συνεργασία στην Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θα ήθελα να ε, χαιρετήσω λοιπόν ε, την νέα νομική βάση, βασισμένη πλέον στη συνθήκη της Λισαβόνας, στην διακυβέρνηση και τα οργανωτικά θέματα, την επεξεργασία πληροφορίας, την ε, λογοδοσία, τη σχέση με ε, τις ε, χώρες, την ανταλλαγή δεδομένων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Όλα αυτά είναι θετικές εξελίξεις. Ωστόσο η ομάδα μου έχει εκφράσει την πρόσφατη απογοήτευσή της σε σχέση με την εντολή της Ευρωπόλ και ζητά τη δημιουργία μιας πραγματικής ε, ερευνητικής ικανότητας στην Ευρώπη. Όπως γνωρίζουμε, ο εισηγητής ζητούσε και εκείνος κάτι τέτοιο, αλλά δυστυχώς τα κράτη-μέλη πολλές φορές έδειξαν διστακτικότητα σχέση με τις διατάξεις που ε, είναι σχετικές με αυτό. Και ο νέος κανονισμός της Ευρωπόλ δεν επέτρεπε την ενσωμάτωση των νέων προκλήσεων σε θέματα ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η έγκριση από κάθε θεσμικό όργανο ε, προτού τις επιθέσεις στον Πατακλάν και στο Σαρλιεμπτό αλλά και πριν τις ε, πρόσφατες επιθέσεις της ε, Βρυξέλλες έχουν δείξει μια ανεπάρκεια. Έχουν δείξει ότι δεν έχουμε λάβει αρκετά στα σοβαρά το έργο μας ως συνομοθέτης. Θα πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένε τροπολογίε που θα αναφέρονται στη θέση του Συμβουλίου και θα αφορούν τρία θέματα. Καταρχά, την εντολή τη Ευρωπόλ γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει η Ευρωπόλη να γίνει ε, κατάλληλη να αντιμετωπίσει τη νέα απειλή στην Ευρώπη. Εάν ε, μείνουν τα πράγματα ε, ως έχει, θα πρέπει να συνεχίσει την αμοιβαία συνεργασία και να ενισχύσει τις ικανότητές της. Την έντολη της Ευρωπόλη όμως αναφέρει ότι κύριος στόχος της είναι η δημιουργία συνεργειών σε ενωσιακό επίπεδο ανάμεσα στις αρχές επιβολής του νόμου και ε, διασυνοριακή συνεργασία για την πρόληψη του σοβαρού εγκλήματος. Έπειτα, η Ευρωπόλ πρέπει να είναι σε θέση να ε, αρχίζει έρευνες και χρειάζονται, χρειάζεται η νομική δυνατότητα που να τη το επιτρέπει. Ε, το υφιστάμενο κείμενο της θέσης του Συμβουλίου δίνει στην Ευρωπόλη τη δυνατότητα να κάνει ένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο αφήνει την απόφαση για το τι θα γίνει στα κράτη-μέλη. Στην ουσία δηλαδή το κάνει προαιρετικό για τα κράτη-μέλη. Έπειτα, επεξεργασία πληροφοριών από τις Εθνικές Μονάδες της Ευρωπόλ. Ο, λόγος τους, ο ρόλος τους θα πρέπει να είναι να διευκολύνουν τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και να δίνουν τη βάση για ε, τις ε, πανευρωπαϊκές έρευνες. Τώρα, σε σχέση με τι ε, πληροφορίε, η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να είναι έργο των εθνικών μονάδων τη Ευρωπόλ, έτσι ώστε να γίνει πραγματικό κόμβος ανταλλαγή πληροφοριών σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε την ε, εξέταση δεύτερη ανάγνωση, τη συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση και δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο όλη τη δουλειά που έχει γίνει ε, και όλες τις μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις μέχρι τώρα έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς μια πραγματικά ολοκληρωμένη αστυνομική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες πολιτικές ομάδες και κάποιοι ε, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν ήδη κάνει έκκληση για καλύτερη αστυνομική συνεργασία και πιστεύω πως εμείς πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Γι' αυτό θα ε, χρειαστούν συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί πραγματικά ένα ισχυρό πλαίσιο. Και φυσικά θα λάβουμε υπόψη τη θέση του Συμβουλίου και τη θέση των άλλων πολιτικών ομάδων για να κοιτάξουμε τι είναι ρεαλιστικό και εφικτό προτού υποβάλουμε τις τροπολογίες μας. Ε, να σας υπενθυμίσω επίσης ότι αυτό που έχουμε ενώπιόν μας είναι μια πραγματική ευκαιρία να ε, ενισχύσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, κάτι το οποίο επιθυμούμε όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Καλώς. Θα ζητήσω από τον εισηγητή στο τέλος να αναφερθεί σε αυτά τα σημεία ιδιαίτερος. Ο κ. Κάρπρος, άλλος ένας και εισηγητής. Για τους πρασίνους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ντία Στεμέρα και τους συναδέλφους. Πολύ καλή δουλειά που έγινε. Χρειάστηκε πολύς χρόνος, σκληρή δουλειά. Έχω τρία σχόλια μας. Πρώτα απ' όλα, εμείς οι πράσινοι έχουμε προβλήματα με τις δυνατότητες που αναφέρονται στο κείμενο, δηλαδή ότι η Ευρωπόλ θα παρέχει πληροφορίες σε ιδιωτικούς φορείς Θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο ζήτημα. Αυτό δεν είναι το καθήκον αστυνομικής υπηρεσίας να δίνει πληροφορίες σε ιδιωτικούς φορείς. Να παραλαμβάνει βεβαίως, αλλά να χορηγεί πληροφορίες όχι. Το πρώτο σχόλιο ήταν αυτό, το δεύτερο. Κάποιος συνάδελφος το ανέφερε. Ο κ. Βάιντενχόλτσα, ο αγαπητός συνάδελφος, είπε ότι έχουμε και την έγκριση του IRU. Ήταν κάτι που αποφασίσαμε ότι θα συμπεριληφθεί σε ξεχωριστό κείμενο για να το εξετάσουμε ξεχωριστά μετά από τις επιθέσεις στο Παρίσι υπήρξε μια γρήγορη αντίδραση, σύμφωνα με την οποία συμπεριλήφθη αυτή η πτυχή στο παλαιό κείμενο. Είχα πει ότι η αντίδραση ήταν πάρα πολύ γρήγορη, υπερβολικά γρήγορη. Έπρεπε να το δούμε ψύχρεμα το σύντημα. Να περιμένουμε να ανακτήσουμε την ψυχραιμία μας μετά από αυτά τα φοβερά συμβάντα Νομίζω με υπεραπλωστευμένο τρόπο συμπεριλήφθη απτυχή και όχι όπως θα έπρεπε. Τρίτον, συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Πέτερσεν. Δεν έχει, επαρκής, δεν έχει δυνατότητες έρευνας η Ευρωπόλ. Θα έπρεπε να έχει όχι μόνο να έχει συντονιστικό ρόλο, να έχει τη δυνατότητα πρωτοβουλίας, να δρομολογεί έρευνες. Συμφωνούμε με αυτό. Θα ήταν καλό να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και θα μπορέσουμε να το εξετάσουμε αυτή την κατάλληλη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που έγινε. Ο κύριος Δίας Δεμέρα πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλό στη συνεργασία μας ακόμα και όταν σε κάποια σημεία διαφωνούσαμε. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πριν ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Δίας μήπως μπορούμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μας βοηθούσε κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Ποιος θα πάρει το λόγο. Ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να είναι άκρως λακωνική και αυτό θα σε ικανοποιεί, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζουμε και όπως ο συγγετής ο κ. Δίας Ντεμέρα υπογράμμισε στην αρχική του παρέμβαση, οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις επί του περιπλόκου αυτού κειμένου χρειάστηκαν χρόνο. Πολύ χρόνο. Το Κοινοβούλιο, υπό την καθοδήγηση του εισηγητού, κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες, ούτως ώστε να διαμορφώσει καταρχάς μια συνενετική λύση στο Κοινοβούλιο με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών ομάδων. Καθώς έγιναν και προσπάθειες να υπάρξει συνεννόηση με το Συμβούλιο πάνω σε αυτό που εμείς θεωρούμε σαν, σαν ένα κείμενο ισορροπημένο και πλήρες. Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο έχει λάβει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσε αυτή η θέση την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου. Και όπως θα διαβάσατε από το έγγραφό μας, θα διαπιστώσατε ότι η άποψή μας είναι ότι οι καθοριστέντες στόχοι της αρχικής μας προτάσεως επετεύθησαν. Θεωρούμε ότι το κείμενο που έχουμε μπροστά μας αφορά μία υπηρεσία η οποία θα ρυθμίζεται, ελπίζουμε, μέσω νομικού εργαλείου που θα ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της συνθήκης της Αβώνας και θα προβλέπει αυξημένη λογοδοσία αλλά και αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στον αφορά τις επιχειρήσεις. Έχοντας αυτό υπόψη, ελπίζουμε ότι οι τελικές φάσεις των μελλοντικών εργάσεων θα ολοκληρωθούν ταχαίως, ούτως ώστε οι νέες διευθετήσεις για τη διακυβέρνηση και τον ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπόλ θα μπορούν να, να υλοποιηθούν. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το Συμβούλιο έχει το λόγο. Ορίστε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω εκ μέρους του Συμβουλίου σήμερα. Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και ο εισηγητής, το Συμβούλιο φρονεί ότι πρόκειται περί καλού αποτελέσματος που πετεύχθη μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων μετά από μακροχρόνιες και δυσχερείς διαπραγματεύσεις. Και το Συμβούλιο πραγματικά θα ήθελε να δει αυτό το σημαντικό νομοθέτημα να εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δίας Δεμέρα, θα επιθυμούσατε να πείτε κάποια λόγια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω επίσης τον εκπρόσωπο της σοσιαλιστικής ομάδας και τον κύριο Κίρκοπ, τον κύριο Πέτερσεν και τον κύριο Τέρι Κάμπρας των Πρασίνων. Ευχαριστώ επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για τα σχόλια τους. Είναι σχόλια τα οποία εμπλουτίζουν το περιεχόμενο και με ενισχύουν έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια μεγάλη συμφωνία σε μια καλή συμφωνία. Σχετικά τώρα με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πέτερσεν θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την εκτίμησή μου για την συνεργασία την οποία είχαμε. να πω ότι συμμερίζομαι τις απόψεις του σχετικά με την πιθανή απόρριψη πιθανώς των τροπολογιών που θα κατατεθούν. Εγώ και η πολιτική μου ομάδα θα καταψηφίσουμε αυτές τις τροπολογίες γιατί οι τροπολογίες αυτές θέτουν εν κινδύνο την διοργανική συμφωνία με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι καλές οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει. Η τροπολογία για την κατάργηση των εθνικών μονάδων δείχνει ότι αγνοούμε τα βασικά θεμέλια της λειτουργίας της Europol. Οι εθνικές μονάδες της Europol είναι θα έλεγα οι κρίκοι οι οποίοι επιτρέπουν στην Europol να λειτουργήσει. Είναι ο διάβλος μέσω του οποίου κυκλοφορεί η ενημέρωση και η πληροφορία και γίνεται επίσης και επεξεργασία της πληροφορίας. Αν δεν υπήρχαν οι εθνικές μονάδες δεν θα υπήρχε η Ευρωπόλ. γιατί οι πηγές τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει θα ήταν ανοιχτές πηγές, ραδιόφωνο, τηλεφωνικές επικοινωνίες, κάτι το οποίο θα ήταν απαράδεκτο λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να υπάρξει επίδειξη κοινή λογικής και γι' αυτό δεν μπορώ να δεχθώ τις τροπολογίες αυτές των φιλελευθέρων. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω α, εκ βάθους καρδίας όλες τις πολιτικές ομάδες που δούλεψαν τόσο και που επέτρεψαν να καταλήξουμε σε αυτή την πρόταση. Καλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα ζητήσω για, από κάποιον άλλον να μιλήσει, θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι δίθεται δύο ζητήματα. Το πρώτο η γενική προσέγγιση και το άλλο είναι το κατά πόσο αποδεκτό, αυτή η προσέγγιση. Δεν θέλω να ξεκινήσω διάλογο τώρα. Δεν νομίζω ότι ήταν επικοδομητικό. Αφήστε με να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ και μετά θα μάθουμε ποια είναι η θέση. Αν αρχίσουμε τώρα δευτερολογίες και μιλήσουν οι φιλελεύθεροι, θα θέλουν και άλλοι να μιλήσουν. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Να ξεκαθαρίσω την άποψή μου. Δύο θέματα τίθενται. Πρώτα απ' όλα γενική προσέγγιση και το δεύτερο είναι κατά πόσο είναι αποδεκτές τροπολογίες. Για τις τροπολογίες είναι δεκτές, ε, θα το εξετάσω βέβαια. Το θέμα της προσέγγισης είναι κάτι διαφορετικό. Συμφωνώ με τη γενική προσέγγιση που ακολούθησε ο εισηγητής και σκιώδης του ECR και των σοσιαλιστών. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις πάμε στη δεύτερη ανάγνωση. Αυτή είναι η θέση που έχω. Θα γίνεται αντιληπτό από τον φιλελεύθερο σκιώδη. Νομίζω ότι το δέχτηκε εξάλλου σε αυτά που είπε. Αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθώ ως Πρόεδρος. Όσον αφορά το παραδεκτόν των ε, τροπολογιών που έθεσε ο κ. Δεμέρα, θα το εξετάσω αυτό δοθέντως το αποτελέσματος τέτοιων τροπολογιών όσον αφορά τη συμφωνία. Θα το εξετάσω αυτό. Θεσμικός πώς. Ε, μου ζητήθηκε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Λοιπόν, δεν έχει νόημα να ξαναπάρει κάποιο το λόγο. Αυτή είναι η θέση μας. Τελικά οι συνάδελφοι μπορούν να τα καταψηφίσουν αυτά. Θα κάνω αυτά τα δύο πράγματα που ανέφερα πριν επανέλθω στο θέμα. ακολουθήσουμε τη γραμμή του εισηγητού και των σκιωδών. 21 Απριλίου είναι η προθεσμία της τροπολογίας και 28 Απριλίου ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ευχαριστώ ξανά τον κύριο Ντίας Δεμέρα και τους σκιώδεις που πήραν το λόγο. Λοιπόν, συνάδελφοι, πάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης ποτέ δεν υπάρχουν εύκολα σημεία στην Επιτροπή μας. Να άλλο ένα σημείο που όπως γνωρίζετε είναι ενδιαφέρον και επίμαχο. Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την όλη κατάσταση και λύσεις όσον αφορά την κατάσταση μη αμοιβαιότητας όσον αφορά τρίτες χώρες για την πολιτική για τις θεωρίες διαβατηρίων. Να επενθυμίσω ότι αυτό αφορά την παρουσίαση ανακοινώσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την όλη κατάσταση και ενδεχόμενε διεξόδου όσον αφορά την ανακοίνωση με τίτλο Ο Μηχανισμό Αμοιβαιότητα που έχει σαν στόχο να εξασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω απολαμβάνουν την ίδια, το ίδιο καθεστώ όσον αφορά τη μην ανάγκη ε, θεωρήσεων. Όταν μια τρίτη χώρα δεν έχει άρρη απέτηση για θεώρηση για κάποιου πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, 24 μήνες μετά τη δημοσίευση της καταστάσεως της μη αβιβαιότητος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να υιοθετήσει κατεξουσιοδότηση πράξης που θα αναστέλει επί 12 μήνων την κατάργηση θεωρήσεως για υπηκόους της χώρας με την οποία η κατάσταση της μη αμοιβαιότητας ισχύει. Ο μηχανισμός επίσης απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συνέπειες της αναστολής της εξαιρέσεως αποθεώρηση για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών μελών αυτής. Σε αυτή την ε, ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι όσον αφορά τον Καναδά και τη ΣΥΠΑ ότι δεν έχει επιτεθεί ακόμα πλήρη αμοιβαιότητα όσον αφορά τι θεωρήσει. Στην παρούσα περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να μην υποβάλει κατεξοδότηση πράξη, αλλά να παρουσιάσει την ανακοίνωση, όπου εκεί καλεί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατεπηγόντω να ξεκινήσουν συζητήσει και να τοποθετηθούν όσον αφορά το επιδεδειγμένο τρόπο πρόοδου από τούτο και στο εξή και να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τι αμοιβέ θέσει του των δύο όχι αργότερα το 12 Ιουλίου του 2016. Θα δώσω το λόγο τώρα λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα μα ενημερώσει για όλε τι εξελίξει και μετά από αυτό θα αρχίσουμε τι συζητήσει, θα ακούσουμε ερωτήσει και σχόλια των μελών. Η Μερίντα Πάικ εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξέρω ότι κάποια μέλη θέλουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα που είναι επίμαχο. Λοιπόν, και πείτε όσοι θέλετε να πάρετε το λόγο. Μπελίντα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή που έθεσε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη μετά από την έγκριση στις 12 Απριλίου της ανακοινώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχα τη δυνατότητα να έρθω σε αυτή την επιτροπή να ενημερώσω για την κατάσταση για την αμοιβότητα των θεωρήσεων τον Δεκέμβριο συνεδρίασή σα. Λοιπόν, να συνοψίσω αυτά που είπατε Λοιπόν, οι αναθεωρημένους μηχανισμούς αμοιβαιότητα των θεωρήσεων ενεκρίθη τον Νοέμβριο του 2013 και σύμφωνα με τον νέο μηχανισμό, αν μετά τις 12 Απριλίου του 2016, δύο χρόνια δηλαδή μετά από τη δημοσίευση των στοιχείων περί υποθέσεων μια αμοιβαιότητας, οι υπόλοιπε τρίτες χώρες που δεν έχουν άρει τις απαιτήσει περί θεωρήσεων για πολίτες ενός ή περισσότερων κρατών μελών, ο μηχανισμός προβλέπει σαν επόμενο βήμα προσωρινή αναστολή της εξαιρε θεωρήσεων για ένα μήνο για πολίτες της τρίτης χώρας, της εν λόγω τρίτης όπως είπατε επίσης, ο κανονισμός απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συνέπειες της αναστολής της εξαιρέσεως της θεωρήσεως για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών μελών αυτής. Η παρούσα κατάσταση έχει ως εξή. Ο Καναδάς εξακολουθεί να εφαρμόζει απέτηση περιθεωρήσεως για τους πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας και είπα απαιτεί θεωρήσεις για τους πολίτες της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πολωνίας και της Ρουμανίας. Επιπλέον, το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε περαιτέρω ταξιδιωτικού ε, ε, περιορισμού το Δεκέμβριο και το ανακοίνωσε αυτό το Δεκέμβριο και αυτό αφορά ενδεχομένω όλα τα κράτη-μέλη που μπαίνουν στο πρόγραμμα εξαιρέσει αποθεωρήσει. Γαλλο... Κάποιο που έχει διπλή υπηκότητα, γαλλική και ιρανική, χρειάζεται θεώρηση τώρα για να πάει στη ΣΥΠΑ. Η ανακοίνωση που θέτει ε, από το Σώμα περιγράφει την κατάσταση λεπτομερώ και αξιολογεί τι πολιτικέ συνέπειε τη αναστολή τη εξαιρέσεω των θεωρήσεων για Καναδά και ΗΠΑ και επίσης καθορίζει την δυνατότητα υλοποίησης αυτού του μηχανισμού. Η ανακοίνωση επίσης αναφέρεται στον Μπρουνέι. Αλλά με τα χαράς λέω ότι το Μπρουνέι κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμως 13 Απριλίου ότι είχε θέσει εξαιρέσεις ε, για αποθεωρήσεις για τους Κροάτες υπηκούς και δίνει παραμονή ανευθεωρήσεων στου στους πολίτες του Λίχτενστάιν. Οπότε πλήρης αμοιβαιότης εξαιρέσεως αποθεωρήσεις με τον Μπρουνάι ε, ισχύει. Ποια είναι τα πορίσματα τότε τη ανακοινώσεω. Καταρχά, όσον αφορά του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, η αναστολή τη εξαιρέσεω θεωρήσει, τουλάχιστον όσον αφορά τι ΗΠΑ, ίσω να έχει αρνητικέ συνέπειε για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Η νομοθεσία των ΗΠΑ προβλέπει ότι θα μπορούσε να απαιτήσει θεωρήσει από του υπηκόου όλων των κρατών μελών, αντί να άρει για του υπηκόου ε, των πέντε κρατών μελών για, τον Καναδά, με βεβαιότητα για την εξαίρεση θεωρήσει δεν είναι κριτήριο όσον αφορά το πλαίσιο της πολιτικής του, οπότε η αντίδραση είναι λιγότερο προβλέψιμη. Δεύτερον, είναι πολύ απίθανο ότι τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να επεξεργαστούν τι αιτήσει για θεωρήσει που θα έχουν αυξηθεί σύμφωνα με τον κώδικα για θεωρήσει, σύμφωνα με του χρονικού περιορισμού που καθορίζονται το σχετικό κώδικα για την έκδοση θεωρήσεω. Θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι έτοιμα να επεξεργαστούν περίπου 10 εκατομμύριο αιτήσει ε, θεωρήσει το χρόνο στη ΣΥΠΑ και 2 εκατομμύρια ε, στον Καναδά να θέσω το πλαίσιο. Σε αυτή τη φάση τα κράτη-μέλη επεξεργάζονται περίπου 120, 120 αιτήσει και στις δύο χώρες ε, αιτήσει θεωρήσεων από πολίτες άλλων χωρών στη ΣΥΠΑ και στον Καναδά. Και το ευρύτερο πλαίσιο ποιο είναι, ότι το 2015 συνολικός αριθμός αιτήσεων Σέγγεν θεωρήσεων σε όλο τον κόσμο ήταν 15,5 εκατομμύρια που επεξεργάστηκαν περίπου 200 προξενικές αρχές, 2.000 προξενίες συγγνώμη. Άρα οι τούντες θα πρέπει να περιμένουν επί μακρόν και να κλείνουν ραντεβού για την αίτηση θεωρήσεως τους. Και θα μπορούμε να υποθέσουμε ότι ενδεχομένω πολλοί από του ετούντε θα αποφασίσουν τελικά να μην έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα καταλήξει σε μείωση στον αριθμό των ταξιδιωτών από Καναδά και ΙΠΑ και θα οδηγήσει σημαντικές οικονομικές απώλειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μείωση 5% είναι συντηρητική εκτίμηση για τον αριθμό τουριστών από ΗΠΑ και Καναδά που θα έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι απώλεια 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για τον τουριστικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αντίκτυπος στις εξωτερικές σχέσεις και στο εμπόριο επίσης θα είναι σημαντικός και το αναφέραμε αυτό στην ανακοίνωσή μας. Ταυτόχρονα, στην ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να παροτρύνει τον Καναδά και τι ΗΠΑ να δείξουν ότι θέλουν τελικά να συμμορφωθούν με την αμοιβαιότητα εξαιρέσει αποθεωρήσει και για τα 28 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτών συγκεκριμένων μέτρων για την επίστευση του σχετικού στόχου. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τον Καναδά, η ανακοίνωση τονίζει τη σημασία ταχεία εφαρμογή της επέκτασης του ETA, δηλαδή ηλεκτρονικής άδειας ταξιδίου, σε συγκεκριμένες κατηγορίες Βουλγάρων και Ρουμάνων ταξιδιωτών. Αυτό όταν εφαρμοστεί θα αναλογούσε στην πράξη σε μια εξαίρεση από θεωρήσεις για περίπου 30% Βουλγάρων και ε, Ρουμάνων ταξιδιωτών. Περαιτέρω, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο Καναδάς θα πρέπει να δερύνει το πεδίο επεκτάσεως του ETA σε άλλου ταξιδιώτες που ταξιδεύουν για πρώτη φορά και αντιπροσωπεύουν χαμηλό κίνδυνο. Γιατί ΣΥΠΑ καλή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΠΑ σαν πρώτο βήμα να προβλέψει ένα μέτρο παρόμοιο με την επέκταση του ETA του Καναδά, δηλαδή ηλεκτρονική έγκριση ταξιδιών, σε ταξιδιώτε με αντιπροσωπικό κίνδυνο. Δηλαδή, είπα να δούνε αν υπάρχει επιλεξιμότητα για έστα για τι πέντε χώρε που αναφέραμε που νόμιμα χρησιμοποίησαν τη θεώρηση την Αμερικανική κατά το παρελθόν. Παραδείγματο χάρη την παρελθούσα δεκαετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί επίση. Είπα να εξετάσουν κάποιε νομοθετικέ ε, Πρωτοβουλίε που προβλήθησαν που θα δώσουν την κατάλληλη ευελιξία στην κυβέρνηση να παρεκκλίνει από το 3% ποσοστό αρνήσεως ε, θεωρήσεων και τα σχετικά κριτήρια ε, και περιορισμό κάποιων ατόμων με διπλή υπηκότητα που περιορίζονται από το να υποφεληθούν από το καθεστώ εξαιρέσεων θεωρήσει. Καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι δυσκολίε που δημιουργούνται για τα κράτη-μέλη λόγω τη αιμονή για απαιτήσει για θεωρήσει για του πολίτε του που ταξιδεύουν στον Καναδά και τι ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να τονίσει ότι αυτές οι ιδέες που αναφέρονται στην ανακοίνωση δεν παρουσιάζονται ως η λύση. Ο στόχος παραμένει εξαίρεση θεωρήσει για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Αυτό είναι αμετάβλητη θέση. Όμως, μία μερική εξαίρεση θεωρήσεων για κάποιες κατηγορίες ταξιδιωτών είναι κάτι καλύτερο από την παρούσα κατάσταση. Εν τέλει, βάσει των αξιολογήσεων για την εφικτότητα και τι διάφορε συνέπειε που υπάρχουν για το εμπόριο, τουρισμό, εξωτερικέ σχέσει, εν γέννη από όλα αυτά, η ανακοίνωση καλεί του συνομοθέτε κατεπηγόντω να ξεκινήσουν συζητήσει και να τοποθετηθούν επί των πιο δεδειγμένων ε, λύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει το ότι η ΛΥΜΠΕ έθεσε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη των εργασιών τη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι όλοι σας ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για αυτό το θέμα και σας απασχολεί ιδιαίτερα. Ε, ο κύριος Δίας Δεμέρα, νομίζω ήταν ο εισηγητής όταν εγκρίναμε την έκθεση σχετικά με τον μηχανισμό αμοιβαιότητας και γι' αυτό θα λάβει το λόγο πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και εσείς είπατε, έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα ιδιαίτερο περίπλοκο. Πριν περάσω στην ουσία της ε, υπόθεσης θα ήθελα να ζητήσω να αναφερθώ στον κανονισμό του 539 σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαιότητας. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε κάποια δεδομένα τα οποία καλό θα είναι να γνωρίζουμε. Μετά από δυόμιση χρόνια διαπραγματεύσεων, οκτώ τριμερείς διαλόγους και οκτώ συναντήσεις σκιωδών καταλήξαμε το Σεπτέμβριο του 2013 με την πλήρη στήριξη του Συμβουλίου και με μεγάλη πλειοψηφία στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατάθεση της νομοθετικής πρότασης έγινε τον Μάιο του 2011. Δεν θέλω να περάσω στις λεπτομέρειες του κανονισμού, αλλά θέλω να θυμίσω ότι ήταν μια διαπραγμάτευση ευρυτάτη. Αξιολογήθηκαν όλα τα θέματα εσωτερικής πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής. Ε, τέθηκε συνολικά το θέμα των θεωρήσεων, του μηχανισμού ε, ανάκλησης των θεωρήσεων όπως επίσης και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κάναμε όλες τις, τις επιμέρους ευαισθησίες και τελικά όμως να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία διασφαλίζει την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των Ευρωπαίων πολιτικών. Αυτό θίγει το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να πούμε εδώ ότι δίδουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διακριτική ευχαίρεια έτσι ώστε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων μηνών μετά την έγκριση του κανονισμού να αναπτύξει τις απαιτούμενες δράσεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρη αμοιβαιότητα. Πέραν όμως αυτού του χρονικού ορίου, όπως είπε και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι σαφές ότι ο κανονισμός ε, είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μία πρόταση για μία κατεξουσιοδότηση πράξη και όχι μία ανακοίνωση. Μία κατεξουσιοδότηση πράξη λοιπόν η οποία έχει σαν στόχο την προσωρινή κατάργηση την έκδοση θεωρήσεων προς τις τρίτες χώρες οι οποίες δεν σέβονται τον κανόνα της αμοιβαιότητας με τα κράτη-μέλη. Το περιθώριο κίνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση μηδενικό και αυτό το επιβεβαίωσε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ένωσης στις 17, 16 μάλλον Ιουνίου του 2015. Ε, Ιουλίου μάλλον του 2015. Δεν θα ήθελα τώρα να μπω στην αξιολόγηση του περιεχομένου αυτής της ενημερωτικής ανακοίνωσης η οποία μας παρουσιάστηκε με αναλυτικό τρόπο από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα πρέπει να συζητήσουμε στην παρούσα φάση τα περί καταλληλότητας ή μη των θεωρήσεων και τις περιπτώσεις του Καναδά, των ΗΠΑ και του Μπρουνέη. Ο κανονισμός στον οποίο αναφερθήκαμε ήδη θέτει ένα συγκεκριμένο όριο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι σαφείς όπως και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Το εδάφιο 3 τι μας λέγει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει με ενεργό τρόπο να επιδιώξει την πλήρη εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας στην έκδοση θεωρήσεων με τρίτες χώρες, συνεισφέροντας έτσι στη βελτίωση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης. Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί λοιπόν με συγκεκριμένο τρόπο και η ουσία είναι στο 1-4-F που λέει ότι αν σε ένα πλαίσιο δύο ετών από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί συγκεκριμένη ανακοίνωση η χώρα για την οποία γίνεται αναφορά δεν έχει καταργήσει την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει μία κατεξουσιοδότηση πράξη για την διακοπή χορήγησης ελεύθερων θεωρήσεων στους πολίτες της συγκεκριμένης τρίτης χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει επίσης μάλλον δεν λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ανακοίνωση γύρω από αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας εξηγήσει βέβαια τι έχει κάνει κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επίτευξης της πλήρους αμοιβαιότητας. Ιδιαίτερα όταν οι συνομοθέτες από την κατάθεση της κατεξουσιοδότησης πράξης και το Συμβούλιο δηλαδή και το Κοινοβούλιο καλούμεθα να συζητήσουμε αν θα την κάνουμε αποδεκτή ή όχι. Αυτή είναι μια δική μας αρμοδιότητα και όχι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντικαταστήσει με μία ανακοίνωση την κατεξουσιοδότηση πράξη. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραβιάσει τον κανονισμό και ιδιαίτερα όταν ε, ο ρόλος ε, της Επιτροπής περιγράφεται με απόλυτο τρόπο από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Να πω ότι εγώ είμαι φίλος του Καναδά, είμαι φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θέλω να υπάρξει επιβολή θεωρήσεων προς τους πολίτες των χωρών αυτών. Αλλά θα ήθελα οι δύο αυτές χώρες να εφαρμόσουν την εξαίρεση στην Πολωνία, την Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Κύπρο και την Κροατία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να πιέσει όσο μπορεί διπλωματικά για να πετύχει κάτι τέτοιο. Πέραν αυτού τίποτα. Πολύ ωραία το θέσατε κύριε Ντίας Δαμέρα. Πρωτού δώσω το λόγο στην κυρία Φαγιόν, θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος να επανέλθει και να μας πει γιατί ε, υπάρχουν οι κατά εξουσιοδότηση στο κανονισμό 539 ε, και τι συμβαίνει με την ε, πρώτερη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Χρειάζεται να ενημερωθούμε και είμαι σίγουρος ότι και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής θα πούν με το δικό τους τρόπο το ίδιο. Η Τάνια Φαγιών έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τον Αγκουστίν. Ήμουν σκιώδη εισηγήτρια το 2013 και αργότερα για τον ίδιο κανονισμό. Και συμμερίζομαι την θέση του και τις ανησυχίες του. Και εγώ θα πω το ίδιο πράγμα με λίγα λόγια. Είναι όντως ένα αρκετά ε, επίμαχο θέμα. Από την άλλη όμως είναι και σαφές ότι το θέμα είναι απλό, ξεκάθαρο. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιο είναι ο κατάλληλος ε, τρόπος για να προχωρήσουμε. Είναι σαφές ότι μετά από μακρές διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτονόητο ε, και άσχετο για μένα στην παρούσα περίπτωση το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σέβεται τον ίδιο του τον κανονισμό δεν είναι αυτό θέμα προς συζήτηση, πιστεύω. Ε, έχει συμβεί πριν από δύο χρόνια και δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει. Σε αυτήν την ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε τρίτες χώρες και σήμερα δεν ακούσαμε ε, καμία αναφορά για την Ιαπωνία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν αναφέρατε σήμερα την περίπτωση της Ιαπωνίας. Μαζί με τη ΣΥΠΑ, τον Καναδά και τον Μπρουνέι, αυτές οι τέσσερις χώρες δεν σέβονται την αμοιβαιότητα ε, για τους ε, πολίτες αυτών των πέντε κρατών μελών της Ένωσης. Κάτι το οποίο τους κάνει πολίτες ε, δεύτερης κατηγορίας και το οποίο θεωρώ απαράδεκτο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρμαχος της ίσης μεταχείρισης όλων των Ευρωπαίων πολιτών Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό 539, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εγκρίνει πράξη κατ' εξουσιοδότηση. Και μετά Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο έχουν τρει μήνες καιρό για να ασκήσουν βέτο εάν έχουν αντίρρηση. Θεωρώ λοιπόν ακατάλληλο να ε, ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας πει τι θα γίνει στη συνέχεια. πρέπει να διαρωτηθούμε αν θα επιτρέψουμε να γίνουν αυτοί οι πολίτες των πέντε χωρών πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ο, μετά, αναφέρατε την τελευταία τροπολογία σχετικά με το πρόγραμμα απαλλαγής αποθεώρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ε, θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες εάν έχουν προηγουμένως ταξιδέψει στο Ιράκ, τη Συρία ή το Σουδάν. Αυτό είναι... Ε, παραβίαση της αρχής της αμοιβαιότητας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα λίγες ε, ακόμα διευκρινήσεις ως προς το τι συμβαίνει εδώ. Και θέλω να ρωτήσω, τι σχεδιάζει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είτε θα εγκρίνετε την πράξη κατά εξουσιοδότηση άμεσα, είτε πρέπει να αλλάξετε τον ίδιο τον κανονισμό σας. Δεν βλέπω άλλη δυνατότητα. Χρειάζονται λοιπόν πιο ξεκαθαρές απαντήσεις από μέρους σας διότι έχουμε διαπραγματευτεί μακρόχρονα και προσφύγαμε στο δικαστήριο και η απόφαση ήταν σαφής για τις πράξεις κατά Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Σεσίλια Γουίξτρομ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά με ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισε να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. η παρούσα ισχύουσα νομοθεσία, έτσι όπως προβλέπετε, έχει ξεκάθαρους κανόνες για την αμοιβαιότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα των θεωρήσεων. Αν δεν εφαρμόσει τη ρύθμιση αυτή, οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν την εφαρμόσουν, τότε θα πρέπει και εμείς να μην την εφαρμόσουμε για τους Αμερικανούς που έρχονται στην Ευρώπη. Οι διακρίσεις εις βάρος των πολιτών Ρουμανίας, Βουλγαρίας και φυσικά όλων των Ευρωπαίων πολιτών με διπλή υπηκότητα είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο και αποτελεί διάκριση. Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι και όπως είπε η κυρία Φαγιόν και οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να διαβουλεύεται με τους νομοθέτες, θα πρέπει απλά να κάνουν αυτό το οποίο τους αναλογεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν σέβονται την αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων και είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μία κατεξουσιοδότηση πράξη η οποία θα διακόπτει την εφαρμογή του προγράμματος κατάργησης των θεωρήσεων με τις ίπα. Τώρα το θέμα είναι γιατί γίνεται η συζήτηση αυτή. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σεβαστεί τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει στα πλαίσια της συνθήκης και του ευρωπαϊκού δικαίου και να παράγει τις πράξεις αυτές όταν είναι απαραίτητο. Αυτή η, η, η επίδειξη υπακοή απέναντι στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι κάτι το οποίο θα χαρακτήριζα απαράδεκτο. Θα πρέπει επίση να ζητήσουμε και από την νομική υπηρεσία να αναφερθεί σε εμά το ταχύτερο δυνατό, στου συντονιστέ, δηλαδή, για οποιαδήποτε μορφή ένομη δράση την οποία θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να αναλάβει αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίσει να αγνοεί τις υποχρεώσεις που έχει εις βάρος του συμφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών. Ή θα είναι λοιπόν μια κατεξουσιοδότηση πράξη ή ένας νέος κανονισμός. Ποια είναι η προοπτική την οποία εσείς επιλέγετε. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταθέσετε μια απλή ανακοίνωση. Πρέπει να αναλάβετε δράση. Thank you. And, uh, Ευχαριστώ. Η Σοφία Ιντεβελτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τα υποθέντα. Εκπλήσωμε, μάλιστα, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παίρνει στα σοβαρά τους Ευρωπαίους πολίτες, πώς μπορεί να περιμένει οι Ευρωπαίοι πολίτες να πάρουν την Κομισιόν στα σοβαρά. Μας εκπλήσει το ότι οι πολίτες είναι απογοητευμένοι στον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπερασπίζεται δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, τότε τι. Τι να περιμένουν πλέον οι πολίτες. Έχετε ένα υπέροχο πρόγραμμα. Έχουμε και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνο για θέσπιση νομοθεσίας και αυτή η θέσπιση νομοθεσίας είναι φρικτή. Ακούγοντας τη διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει Κοιτάξτε, θα καλέσουμε τη ΣΥΠΑ. Ε, αν θα είχαν την καλοσύνη, του παρακαλούμε, θερμοπαρακαλούμε να αντιμετωπίζουν αξιοπρεπώ πολίτε μα. Όχι, δεν καλούμε τις ΣΥΠΑ. Περιμένουμε, είπα, να συμπεριθούμε τρόπο. Είναι εταίροι. Απαιτούμε, περιμένουμε να αντιμετωπιστούν οι πολίτες με εξωπρεπή τρόπο. Απηχώ και τα όσα είπε η συνάδελφός μου η Σεσίλια Βίξτρομ. Αυτό το κοινοβούλιο τώρα θα πρέπει να βρει τρόπους ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της. Ίσως αυτό να συνεπάγεται και ε, προσφυγή στα δικαστήρια κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μη δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως θα έπρεπε. Και τέλος αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι το πρόγραμμα εξαιρέσεω αποθεωρής των ΗΠΑ χρησιμοποιείται πολύ συχνά από τις ΗΠΑ για να εκβιάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να λαμβάνει διάφορα μέτρα ασφαλεία η Ευρωπαϊκή Ένωση αν αυτό το πρόγραμμα εξαιρέσει αποθεωρήσει χρησιμοποιείται ότι ο τρόπο, αλλά δεν καλύπτει καν όλου του πολίτε Ευρωπαϊκή Ενώσεω και υποκλίνεται προ τη ΣΥΠΑ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε τι. Και ζητάει και συγγνώμη που ενοχλεί τη ΣΥΠΑ, τι να πω, ένα απαράδεκτο. Όλοι οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και όλα τα κράτη μέλη Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Και περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σέβεται αυτή την αρχή εξίσου. Ψηφίσαμε εδώ και δύο χρόνια. Στηρίζοντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει τα αποτελέσματα, τα αναμενόμενα. Είδε μη το Κοινοβούλιο σε κάποια φάση θα εκφράσει την απώλεια εμπιστοσύνη τη, απώλεια τη εμπιστοσύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι θα πούμε αυτά που θέλουμε με τον αμήμητο τρόπο μα, όπω έλεγα. Λέει ο Πρόεδρο, ο κ. Πάβελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να είμαι πολύ σύντομο και να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει κατά πόσο ζήτησε να μάθει από τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά κατά πόσο ζήτησαν ε, να είπα και ο Καναδάς να υπολογίσει ποιες είναι οι συνέπειες που απαιτούν θεωρήσεις από πολίτες κάποιων χωρών. 20 εκατομμύρια Ρουμάνοι δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα 26 κράτη-μέλη όσον αφορά τον Καναδά και 23 άλλα κράτη-μέλη όσον αφορά τις ΣΥΠΑ. Στέλνουμε προς υπάρχουν προτάσεις κάτι να γίνει, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Ίσως μπορεί να υπάρχει μερική εξαίρεση από θεωρήσεις, κάτι είναι αυτό, αλλά όχι αρκετό. Αισθανόμαστε σαν πολίτε δεύτερη κατηγορία. Η Ρουμανία κατονομάζεται από τη ΣΥΠΑ σαν στατηγικός εταίρο για τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά δεν καλύπτονται οι πολίτε μα από την εξαίρεση αποθεωρήσει. Μα ζητούν να κάνουμε πράγματα για να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και του ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά είμαστε πολίτε δεύτερη κατηγορία. Επί 10 χρόνια περίπου είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, αλλά ακόμα αισθανόμαστε σαν να μην είμαστε εδώ. Δεν είμαστε στο Σέγγεν. Δεν μας καλύπτει και το σύστημα εξαιρέσεων που Περιμένουμε αλληλεγγύη από τους πολίτες των χωρών όσον αφορά την κρίση Μα ζητούν αλληλεγγύη για τα προβλήματα των προσφύγων, αλλά από την άλλη πλευρά δεν δέχομαστε εμεί υποστήριξη προβλήματα που έχουμε εμεί. Ευχαριστώ πολύ, και Στίβενς έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, όλοι α, γνωρίζουν ότι η τουριστική βιομηχανία από τη Βόρεια Αμερική, οι τουρίστες από τη Βόρεια Αμερική παράγουν 60 εκατομμύρια. Ε, αντιστοιχούν στα έσοδα από την αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι ο τουρισμός από τη Βόρεια Αμερική και πόσο εξαρτώμεθα από αυτό. Ε, χαιρόμαστε διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την απόφαση επιτρίμηνο για αυτό το σημαντικό θέμα διότι δίνει έτσι το χρόνο σε όλα τα μέρη να καταλήξει καλή συμφωνία. Λαμβάνοντα υπόψη τις επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες πλήττεται η οικονομία μας. Ξενοδοχεία και εστιατόρια πλήττονται. Χρειαζόμαστε πραγματικά τουρίστες. να απαιτούνται θεωρήσεις από τους τουρίστες που θέλουν να έρθουν από Καναδά και τη ΣΥΠΑ είναι κάτι που θα μειώσει τη ροή την τουριστική. Απευθύνω έκκληση σε όλα τα μέρη προς κατανόηση και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ε, καλή συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σίπελ. Thanks a lot. Σας ευχαριστώ πολύ. Μοιράζομαι και εγώ τις απόψεις πολλών ε, που μου μίλησαν πριν από μένα και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε η Σοφίν Φέλντ, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κάνει κακή νομοθεσία. Όχι, δεν είναι αυτό. Αρνείται να νομοθετήσει, αρνείται να λάβει μια σαφή θέση και αρνείται να αναλάβει ευθύνες. Αυτό όμως είναι, και το, είναι, είναι το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το μόνο θεσμικό όργανο που μπορεί να κάνει νομοθετικές προτάσεις και αν καταλαβαίνω καλά τη διαδικασία είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν μια πράξη κατά εξουσιοδότηση. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, εάν δεν ήταν η Κύπρος, η Βουλγαρία, η η Ρουμανία, αλλά μετά τις επιθέσεις η Γαλλία ή το Βέλγιο, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν η ίδια. Δεν νομίζω. Γι' αυτό αναμένω μια σαφή απάντηση. Θα ήθελα οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι υπόλοιπε χώρε να ε, εργαστούν πάνω στην αμοιβαιότητα των θεωρήσεων και θα ήθελα να δω και ανάληψη ευθύνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι με αυτόν τον τρόπο κάθε άλλο παρά αυτό δείχνει ορισμένοι από τους πολίτες μας, όπως οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Κύπροι και άλλοι, δεν μπορούν να ταξιδέψουν ε, απαλλαγμένοι από την υποχρέωση θεώρησης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κάποιοι άλλοι πολίτες πριν από μερικά χρόνια ε, δεν επιτρέπεται δεν ε, επιτρεπόταν να ταξιδέψουν χωρίς θεώρηση. Αυτό γινόταν όμως παλιά και εγώ προσωπικά ξέρω αρκετούς πολίτες, γερμανούς πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς θεώρηση στις ΗΠΑ Πολιτείες και δεν μπορούν να επισκεφτούν τις οικογένειές τους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ επιθυμώ μία ξεκάθαρη απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να διασφαλιστεί αμοιβαιότητα των θεωρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ράντεφ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 10 χρόνια και μας θυμίζουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δυστυχώς πως δεν είμαστε πλήρε μέλος ακόμα. Η επέκταση του καθεστώτος για τις θεωρήσεις για τους βούλγαρου πολίτες που ταξιδεύουν στον Καναδά και τις ΗΠΑ είναι ένα ακόμα παράδειγμα γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση πρέπει να δείξει αλληλεγγύη και να το αποδείξει η κυβέρνηση του Καναδά πρέπει να διευκολύνει ε, τις, ε, την, ε, την απαλλαγή θεωρήσεων για τους βούλγαρους πολίτες και ελπίζω αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Ελπίζουμε επίσης οι Ηνωμένε Πολιτείες να ακολουθήσουν ε, αυτό το δρόμο σε σχέση με την απαλλαγή από θεώρηση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι τα μέτρα που θέλει να ε, λάβει για να συνεχίσει ο διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά έτσι ώστε να απαλλαγούν από την υποχρέωση θεώρησης οι Βούλγαροι πολίτες και οι πολίτες των υπόλοιπων κρατών μελών που πλήττονται από αυτό το μέτρο. Τον ε, Απρίλιο παραπέμπτηκε το θέμα ε, αυτό εξαιτίας της παραβίασης του ε, κανονισμού. Ελπίζω ο κανονισμός αυτός να εφαρμοστεί στην ολότητά του χωρίς παραπάνω καθυστερήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χολμάρη έχει το λόγο. Και εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, είναι πιο συνεπής στις ενέργειές της. Πάρα πολύ καιρό ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι ανοιχτά ε, αυτά τα έγγραφα για μένα δεν έχει καμία λογική ορισμένοι να είναι απαλλαγμένοι από την υποχρέωση θεώρησης και ορισμένοι όχι. Για μένα δεν, υπάρχει, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αμοιβαιότητα σε ορισμένες περιπτώσεις και σε άλλες ε, όχι. Γιατί πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα, δεν ξέρω, στην Ουγγαρία ή στην ε, Γερμανία. Εάν υπάρχουν φόβοι για... Ε, εγκληματίες οι οποίοι μπορεί να εισέλθουν στο έδαφος των ΗΠΑ ή του Καναδά μπορούν να ε, αναλάβουν άλλη δράση. Ε, διότι, ξέρετε, οι διαρρήκτες δεν χρειάζονται, δεν περιμένουν πρώτα να πάρουν βίζα για να κάνουν ένα έγκλημα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, υπάρχουν πλαστές ε, ταυτότητες, πλαστά διαβατήρια, πλαστές θεωρήσεις. Οι εγκληματίες θα βρουν τρόπο να μπουν στις χώρες αν θέλουν. Και πιστεύω πως η υποχρέωση, η άρνηση μάλλον για την απαλλαγή από θεωρήσεις είναι το μικρότερο ε, πρόβλημα που θα τους ε, δημιουργηθεί. αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξει επιτέλους μια συμφωνία. Γι' αυτό όμως χρειάζεται και βούληση. Έτσι απλά μια άρνηση και απραξία για μένα είναι απολύτως απαράδεκτο. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ενωμένο στην άποψή του, διότι με αυτόν τον τρόπο στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άκουσα πολύ προσεκτικά, προσπάθησα να καταλάβω τι συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Τι πέτυχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις. Το μόνο που κατάλαβα είναι κάτι αρκετά κοινικό από πλευρά Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν παραβιάσουμε κάτι από τις σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά, θα υποστούμε απώλειες σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει οι πήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάθονται στη σειρά ε, για θεωρήσεις κάποιων χωρών. Τι γίνεται, τι βήματα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άρση της απαιτήσεως για θεωρήσεις για τους πολίτες κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βλέπω λύση. Τι περιμένετε από εμά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι βήματα θα κάνετε εσείς Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επόμενους μήνες, ούτω ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία που έχετε εσείς εγκρίνει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα επανέλθω στην Πελίντα Πάικ, που ήρθε αναμένοντας αυτά που άκουσε, πιστεύω. Αυτά που είπαν οι βουλευτές. Στην απάντησή σας θα θέλαμε να ακούσουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εφαρμόζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό εξόργησε τα μέλη όλων των πολιτικών ομάδων. Γιατί δεν εφαρμόστηκε ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η κατεξουσιοδότηση πράξη που εκπονήσατε. Θέλουμε απάντηση. Υποψιαζόμαστε ποια είναι η απάντηση, θέλουμε να την ακούσουμε όμως. Έχουν τεθεί και άλλες ερωτήσεις. Δημιουργεί οργή το θέμα. Συζητούν οι συντονιστές για το ποια δράση μπορούμε να εφαρμόσουμε. Το βασικό ερώτημα απαντήστε, αν έχετε την καλοσύνη, τώρα που θα πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω πράγματι να το κάνω αυτό. Το ιστορικό, το υπόβαθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και όλοι στο Κοινοβούλιο, φρονεί ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης αμοιβαιότητα της θεωρήσης. Μα ρωτήσατε τι κάναμε. Προσπαθούσαμε. Συζητούσαμε με τις ανλογοχώρες τα τελευταία δύο χρόνια. Σε ανακοινώσεις ενημερώσαμε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα τεκτενόμενα. Εξηγήσαμε τη διαδικασία. Σας την εξηγήσαμε. Κοιτάζοντα προ το παρελθόν, την τελευταία δεκαετία, το 2005, 18 κράτη-μέλη ή συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν μας κοινοποίησαν ότι υπήρχαν οκτώ τρίτες χώρες που απαιτούσαν θεωρήσεις από τους υπηκούς τους. Δυστυχώς έχουμε πέντε κράτη-μέλη που πλήττονται από απαιτήσεις για θεωρήσεις από δύο τρίτες χώρες, αλλά νομίζω ότι πετύχαμε πρόοδο όσον αφορά την αμοιβαιότητα για θεωρήσεις. Μην το λησμονούμε. Όσον αφορά την Ιαπωνία, που έθεσε η Τάνια Φαγιόν. Η Ιαπωνία έχει επεκτείνει την εξαίσθηση θεωρήσεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου για Ρουμάνους υπηκόους Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα αμοιβαιότητας με την Ιαπωνία. Οι Ρουμάνοι ελεύθερα πάνε στην Ιαπωνία χωρίς θεώρηση. Συνεχώς παρακολουθούμε την κατάσταση. Και περιμένουμε το καθεστώς να επεκταθεί πέραν της 31 Δεκεμβρίου του 2018. Δεν υπάρχει πρόβλημα την Ιαπωνία όσον αφορά μία αμοιβαιότητα. Σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί Χρησιμοποιούμε όλε τι επαφέ σε όλα τα επίπεδα, στι συνομιλίε με τι κυβερνήσει ΗΠΑ και Καναδά. Και χαίρομαι που βλέπω ότι υπάρχουν και αξιωματούχοι παρόντε των ΗΠΑ και του Καναδά στη συνεδρίαση και θα διαβιβάσουν τα μήνυματά μα, τα μήνυματα του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνομίλησε με του ομολόγου τη την περασμένη εβδομάδα και θα λάβουν χώρα και άλλε επαφέ υψηλού επίπεδου τι επόμενε εβδομάδε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υποβάλει πράξη σε αυτή τη φάση. Είναι σαφή η νομοθεσία, πράγματι. Η Σόφι Ινφελτ αναφέρθηκε σε καλύτερη νομοθεσία. Πράγματι, καλύτερη νομοθεσία, βλέποντας τη διοργανική συμφωνία, απαιτεί από εμά να διαβουλευτούμε του εμπλεκόμενου φορεί την προετοιμασία τη κατεξουσιοδότηση πράξεω. Άρα, μια κατεξοδότηση πράξη δεν μπορεί να υποβληθεί χωρί να γίνει κατάλληλη προετοιμασία. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να τοποθετηθούν επ' αυτού του ζητήματο. Η νομοθεσία προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάλει κατεξοδότηση εν πράξη, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο να μπλοκάρει την ελόγω πράξη. Κάποιο από εσά μπορεί να δράσει μονομερό και τα δύο θεσμικά όργανα εκπροσωπούνται εδώ και τα δύο θεσμικά όργανα εκπροσωπούνται εδώ σήμερα. Θεωρούμε ότι είναι λογικό να διεξαχθεί τώρα η συζήτηση αυτή το επόμενο τρίμηνο. Είναι σημαντικό να διευθετηθεί το πρόβλημα και γι' αυτό σας καλούμε να εκφραστείτε επί της ουσίας. Κατανοούμε τις απόψεις που έχετε περί νομοθεσίας, γνωρίζουμε τι λέει η νομοθεσία. Θέλουμε να ξέρουμε ποιες είναι οι απόψεις σας για την περαιτέρω πρόοδο. Σας δώσαμε την αρχική αξιολόγηση των συνεπειών που είναι σημαντικές. Συμφωνούμε ότι είναι απαράδεκτο να εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, τρίτες χώρες να επιβάλλουν θεωρήσεις επί κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσης όταν δεν απαιτούμε θεωρήσεις για επικούς αυτών των τρίτων χωρών. Όπως είπατε στην αρχή Πρόεδρε, πρόκειται περί επιμάχου και δυσκόλου ζητήματο, το δεχόμαστε και θέλουμε διάλογο μαζί σας και με το Συμβούλιο, η Προεδρία εκπροσωπείται εδώ, θα θέλαμε αυτό να γίνει το επόμενο τρίμηνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν μεταξύ μας διαφορές. Είμαστε ξεκάθαροι σε σχέση με το επιθυμούμε. Θεωρούμε ότι δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο, δεν εκδίδεται την κατεξουσιοδότηση πράξη, είναι σαφής η αντίληψή μας, δεν είναι δικό μας καθήκον να συζητήσουμε το τι μπορεί να γίνει. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε πρέπει να το κάνετε και σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Σόφι, διαδικαστικό ή θες κάτι άλλο να προσθέσεις. Η Επιτροπή, Επιτροπή αυτό το οποίο λέει είναι ότι κοιτάξτε πρώτα εμείς πρέπει να διαβιλευτούμε. Λοιπόν, αφού ακούσατε τη συζήτηση που προηγήθηκε, κατέστη σαφές ότι υπάρχει μια ευρυτάτη ε, συμφωνία για τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Οπότε τώρα θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να καταθέσετε αυτή την πράξη. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Κοιτάξτε, είναι το μοναδικό πιθανό συμπέρασμα από αυτά που είπα. Δεν ξέρω τι είχε στο νου σου όταν μίλαγε η Επιτροπή, αλλά πάντως ε, η ερμηνεία αυτών που είπε δεν είναι η ίδια η δική μου και η δική σου. Δεν το είπε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να, πούμε ευχαριστούμε λοιπόν την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω μαζί σας, αυτό δεν είναι αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνώ με τη Σόφη ότι αυτό θα έπρεπε να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, λέει ο κύριος Μωράες. Ξέρουμε τι θα έπρεπε να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλετε μπορούμε να πιούμε ένα καφεδάκι και να τα συζητήσουμε όλα αυτά μεταξύ μας. Αλλά θα πρέπει οι συζητήσεις αυτές να τηρούν κάποιους κανόνες, παρακαλώ απαιτείται μια κάποια τυπικότητα στις ε, ανταλλαγές απόψεων. Λοιπόν, συμφωνούμε χωρίς καμία διαφορά μεταξύ μας. Το θέμα θα το συζητήσουν οι συντονιστές έτσι ώστε για τα μέλη ιδιαίτερα που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες το θέμα παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα πρέπει να κάνουν κάποιο πρόγραμμα δράσης οι συντονιστές. Ευχαριστώ ξανά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσία της και συνεχίζουμε. Περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Ψυχοτρόπες ουσίες λοιπόν και μέτρα ελέγχου στις 7 Απριλίου το EMCDDA και η Europol παρουσίασαν τη δεύτερη έκθεσή τους για την αγορά ναρκωτικών στη Λίμπε. Ενημερωθήκαμε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν πάνω από 560 ψυχοτρόπες ουσίες το Συμβούλιο έθεσε χρονική προθεσμία τριών μηνών για την έκδοση γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες. Γι' αυτό λοιπόν, για να ακούσουμε περισσότερα στοιχεία, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μπόνι. Κύριε Μπόνι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Θα ήθελα σύντομα να παρουσιάσω την ακθεσή μου για την εφαρμοστική απόφαση για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες την φλάκα, γκράβελ ή εν περιπτώσει ουσίες που ε, αποτελούνται κυρίως από πυρολιδίνη. Έχει αξιολογηθεί η ουσία αυτή από την Επιστημονική Επιτροπή της EMCDDA και τα ευρήματα έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 27 Νοεμβρίου του 2015. Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης στην ουσία λέγουν ότι η ουσία αυτή ε, είναι μια ισχυρή ψυχοτρόπος ουσία, υπάρχει και στις 28 ε, χώρες και στην Ορβηγία και στην Τουρκία και εισάγεται η βασική ουσία κυρίως από την Κίνα έχουν υπάρξει 115 θάνατοι και 191 σοβαρές τοξικές δηλητηριάσεις σε 8 κράτη-μέλη. Και δεν έχει καθοριστεί η ιατρική χρήση της ουσίας αυτής στην Ένωση. Η χρήση της ξεκίνησε στην αρχή του 21ου αιώνα και δεν περιλαμβάνεται στον, έλεγχο των, στον κατάλογο των υποέλεγχο ουσιών της Σύμβασης ε, των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και της Σύμβασης του 1971 των Ηνωμένων Εθνών για τις ψυχοτρόπες ουσίες. Δεν ε, είναι υποαξιολόγηση και δεν παρακολουθείται από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών που είναι προϋπόθεση για να υπάρξει μια ρύθμιση σε επίπεδο ευρωπαϊκού ε, συστήματος. Μιας και είναι επικίνδυνη σύμφωνα με την αξιολόγηση της EMCDDD μπορεί να προκαλέσει delirium και γι' αυτό υπάρχουν μέτρα τα οποία θα πρέπει να γίνουν Πρέπει λοιπόν να κάνουμε δεκτή την πρόταση γύρω από την πυρολιδίνη. Σας ευχαριστώ κύριε Μπόνη. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το θέμα και ξέρω πως ενδιαφέρει όλους εμάς. Θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές με τη σειρά και θα αρχίσω με την Άννα Χέντ. Θα θέλατε το λόγο? Ε, συνάδελφοι, συνάδελφοι, θα ζητήσω συγγνώμη. Ποιος θέλει το λόγο. Δεν υπάρχει κατάλογος ομιλητών. Εντάξει, δεν θέλω να σας ε, βάλω να μιλήσετε με το ζόρι. Αν θέλετε, μιλήστε. Κύριε Μπόνη, στις 25 Απριλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροπολογιών. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι. Ναι, θα περιμένω τις τροπολογίες, αλλά πιστεύω ότι μετά από την ανάλυση της MCDDA ε, το θέμα είναι σαφές. Θα συνεχίσουμε όπως έχουμε προγραμματίσει. Μάλιστα. Ε, Εξαρτόμαστε από σας γιατί ξέρουμε πώς θα τα καταφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης. Και θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη και για την καθυστέρηση. Ε, Όμω ε, χαίρομαι που επιτέλου καταφέραμε να βάλουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αναφέρομαι στην αποστολή στην Τουρκία από τι 8 έω 11 Φεβρουαρίου. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, ε, που καταφέραμε να στείλουμε μια αποστολή στην Τουρκία για την κατάσταση με τους πρόσφυγες. Θα δώσω λοιπόν ευθύ αμέσω το λόγο στην Σιλβί Γκυγιό, με επικεφαλής της αποστολής, που θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεση σχετικά με την αποστολή. Και μετά θα λάβουν το λόγο τα μέλη που το επιθυμούν. Σιλβί, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, έχουμε ελάχιστο χρόνο, θα προσπαθήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε πλήρως, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, Έχω μια έκθεση πληρέστατη που συνετάχθη. Ευχαριστώ τα μέλη που συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή. Πιστεύω ότι το, η όλη ατμόσφαιρα ήταν ε, ευχάριστη και συμπαθής. Ευχαριστώ και το προσωπικό της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που ήρθε μαζί μας και κυρίως την Καρτίν Λιμπέρ που είναι εδώ και τον Νίκολα η Κατρίν ήταν πολύ ακριβής όσον αφορά το συντονισμό των κινήσεων χρονικά και την ευχαριστώ για τη συμβολή της. Ευχαριστώ και την ομάδα των διερμηνέων που ήταν και των μεταφραστών και τους υπεύθυνους στην επικοινωνία. Πήγαμε στην αποστολή αυτή την ιστορική στιγμή που θα έλεγα που λάμβαναν χώρα βομβαρδισμοί επί του Χαλεπιού οπότε καταφθάναν πρόσφυγες στα σύνορα με την Τουρκία ε, και είχαν ανοίξει τα σύνορα πριν τη συμφωνία βέβαια Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ενώσεως που συνήφθη τότε. Τρεις μέρες είμαστε στην αποστολή. Το πρόγραμμα ήταν πολύ φορτωμένο. Αναφέρω και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Άγκυρα που μας βοήθησε πολύ Πήγαμε σε επιτόπιες επισκέψεις και ήρθαμε σε επαφή με διαφόρους εμπλεκομένους φορείς, αξιωματούχους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ε, η επίσκεψη στο, στα τόπεδα εκεί πέρα, στις, στους καταβλισμούς, ε, στις... Ε, πήγαμε λοιπόν, είδαμε και τις σκηνές και τα, αυτούς που μένανε και στα κοντέινερ Επισκεφθήκαμε και οικογένειε προσφύγων εκτός των καταβλισμών. 89% ε, από αυτούς είναι πρόσφυγες εκτό των οργανωμένων καταβλισμών που έχουν οργανώσει οι Τούρκοι. Είναι άνθρωποι ε, που περνούν πολύ δύσκολα. Θα επανέλθω σε αυτό. Ήρθαμε σε επαφή με ΜΚΟ επιτόπου χωρίς να μιλήσω με τους διάφορους εθνικούς φορείς εκπροσώπους τη τοπική αυτοδιοίκηση με του οποίου θα σε επαφή. Αυτοί που ενδιαφέρονται τις λεπτομέρειες μπορούν να εξετάσουν τα γραφόμενα. Λοιπόν, κάποιες εκτιμήσεις. Η έκθεση αναφέρει ότι η κατάσταση όσον αφορά τη σύγκρουση ε, είναι κάτι που, ε, να σταματήσει η σύγκρουση είναι κάτι που θα βελτιώσει την επιτόπια κατάσταση, ξυπακούεται. Σημειώνουμε τις προσπάθειες των τουρκικών αρχών που προσπαθούν παντιοτρόπως να δεχτούν τους Σύρους πρόσφυγες στην επικράτεια της χώρας και γίνεται σημαντική προσπάθεια που έχει συνέπειες όσον αφορά τους ντόπιου κατοίκους και τις τοπικές κοινότητες χρειάζεται πιο στενή συνεργασία από ό,τι κατά το παρελθόν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Τουρκίας. Αυτή η έκθεση δέχεται όμως ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των προσφύγων δεν είναι στους καταβλισμούς και πιστεύω ότι απαιτεί αποφασιστική υποστήριξη για να βγουν, να υπάρξει καλύτερη στέγαση, διατροφή, ε, παιδεία για τα παιδιά και πρόσβαση στην ε, απασχόληση. Ε, και είναι συγκινητική κατάσταση που αντιμετωπίζουν και τα προβλήματα. Αναφέρεται στην έκθεση ότι τα 3 δισεκατομμύρια που έγιναν 6 δις έκτοτε που δίδονται στην Τουρκία θα πρέπει να προσανατολιστούν προς την τοπική αυτοδίκηση Τουρκίας και τους ΜΚΟ, τους επιτόπιους ΜΚΟ και να υπάρχει παρακολούθηση το πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται. Θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε η οικονομική υποστήριξη κυρίως προς το World Food Program και την είπατε αμοστία του ΟΗΕ είναι απαραίτητα στοιχεία διότι εκεί που ήμασταν οι πόροι προς, μειωνότανε προς αυτούς τους φορείς και αυτό επηρέαζε άμεσα την ζωή των προσφύγων επιτόπου. Νομίζω ότι κάπως ρυθμίστηκαν έκτοτε τα πράγματα και είπαμε ότι χρειάζεται υποστήριξη της μεταεγκατάστασης ακόμα και αν αυτή για την ώρα δεν ε, φαίνεται να λαμβάνει χώρα και να προσπαθούν ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη να το πραγματοποιήσουν αυτό. Συνοπτικά είναι τα σχόλια. Είναι πολύ πυκνή βλέπετε η έκθεση. Εγώ ε, είμαστε ανοιχτοί όσον αφορά τα σχόλια των άλλων μέλων της αποστολής, όπως της Άννα Μαρία. Και τα όσα υπόθηκαν στον αφορά και δραστηριότητα της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Εν συντομία λοιπόν αυτά έχω να πω για την αποστολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γκυγιόμ. Όπως είπατε η Άννα Μαρία και η Τάνια Φαγιών θέλουν να λάβουν το λόγο. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι, μάλιστα. Κλείνω λοιπόν τον κατάλογο των ομιλητών. Άννα Μαρία, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την ε, Σιλβή για την ε, καλή συνεργασία, αλλά και το επιτελείο της, ε, που μας συνόδευσε στην αποστολή. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική αποστολή και συμμερίζομαι και εγώ τα ίδια συμπεράσματα της έκθεσης που θεωρώ πως είναι πολύ καλή πιστεύω πως πρέπει να αναγνωρίσουμε την τεράστια προσπάθεια που έχουν καταβάλει οι τουρκικές αρχές για να φιλοξενήσουν με αξιοπρέπεια 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Χρειάζονται να γίνουν περισσότερα ε, στην ε, ε, Τουρκία για να διανεμηθούν τα κονδύλια με το σωστό τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, ήμουν η μόνη Ευρωβουλευτή παρούσα στην αποστολή στην Άγκυρα και θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω και δύο ακόμα στοιχεία τα οποία θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικά για το αποτέλεσμα των συναντήσεων. Το πρώτο ήδη καλύπτεται από την έκθεση και είναι η εστίαση στην επαναγκατάσταση. Αυτό ήταν και ε, κύριο θέμα για την αρμοστία. Η επαναγκατάσταση είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να εισέλθει κανείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, αυτή τη στιγμή οι καθυστερήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που συζητήθηκε και προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη με την επανεγκατάσταση. Όταν μιλάμε δηλαδή για νόμιμους ε, τρόπου εισόδου, αυτός είναι ο κυριότερος. Έπειτα, το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι η πληροφόρηση. Εντοπίσαμε ε, ότι μέσω του ε, ΑΣΑΜ, που είναι η μεγαλύτερη ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στην περιοχή ότι υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις στην καταγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων των ε, ε, προσφύγων. Το σύστημα αυτό είναι πάρα πολύ καλό αλλά αυτό που κάνει η Πατιαρμοστία είναι το εξή. Προσπαθεί μαζί με την Τουρκία να δημιουργήσει μια κοινή βάση δεδομένων που θα βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και έτσι θα δημιουργήσει ικανότητε ε, που θα δώσει η Πατιαρμοστία στην Τουρκία έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια εναρμονισμένη βάση δεδομένων. Πιστεύω πως πρέπει να δούμε με ποιους τρόπους θα δημιουργήσουμε πρότυπα, θα δημιουργήσουμε μεθοδολογία που θα είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, την καταγραφή. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και εμείς πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Δηλαδή, οι πρόσφυγες που φτάνουν από την Τουρκία στην Ελλάδα, τι γίνεται, από, καταγράφονται από το σύστημα της Τουρκίας ή όχι, διαγράφονται από αυτό. Όταν φτάνουν στην Ελλάδα μπορούμε με κάποιο τρόπο να δημιουργήσουμε κάποιο σύστημα μηδέας αναγνώρισης και διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Εντάξει, δεν πρέπει να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία. Διότι πιστεύω πω θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε σε αυτό. Όταν οι πρόσφυγε φτάνουν στην Ελλάδα, αρχίζουμε από το μηδέν. Και ε, πιστεύω πως ένα τέτοιο σύστημα θα, προσπαθ, μας βοηθούσε να καταπολεμήσουμε την παράνομη είσοδο και να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε τη διαδικασία ε, νόμιμης εισόδου. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως ε, αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο ε, κείμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Τάνια Φαγιών έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω την Σιλβή, η οποία ήταν εξαιρετική στην ιδιότητά της ως πρόεδρος. Να ευχαριστήσω επίσης και όλο το επιτελείο που μας συνόδευσε στην αποστολή. Τώρα, στην αποστολή μας φυσικά είδαμε την καλή πλευρά της ε, πραγματικότητας, την, ε, τις καλές περιπτώσεις, γιατί στη Καζιαντέπ τα, οι, οι καταβλισμοί υποδοχή είχαν κατασκευαστεί για τις πιο βάλλοντες ομάδες και η οργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή. Όμως, ε, όπως θα διαβάσετε και στην έκθεση, μιλάμε για το 10-20% ε, των προσφύγων που φιλοξενούνται σε, αυτά τα, σε αυτές τις εγκαταστάσεις στην Τουρκία. Οι υπόλοιποι βρίσκονται στον δρόμο. Το να κάνουμε λόγο για αυτήν την κατάσταση στην Τουρκία, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι τουρκικέ αρχέ κάνουν ό,τι μπορούν. Όταν όμω ε, συζητήσαμε μαζί του, κατέστησα σαφέ ότι τα τελευταία πέντε χρόνια δεν κάνουμε και πολλά για να του βοηθήσουμε. Εγώ προσωπικά εξεπλάγει, σοκαρίστηκα σχεδόν με αυτά που άκουσα. Αν δεν κάνω λάθος, ε, συνομίλησα με τον Υφυπουργό Εσωτερικών τη Τουρκία και τον ε, τον ρώτησα ε, τι συμβαίνει σε μια περίοδο που ήταν κλειστά τα σύνορα με τη Συρία και περίμενα κόσμος να μπει στην Τουρκία. Τον ρώτησα λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε αν ε, κολλήσουν εκεί οι άνθρωποι. Και τι, ξέρετε τι μου είπε, δεν είναι δικό μας το πρόβλημα, πάρτε τους αν τους θέλετε. Ήταν πολύ σκληρή δηλαδή αυτή η δήλωση, πολύ σκληρά τα λόγια του και εγώ προσωπικά είδα έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ε, Τουρκία και την Ευρώπη, μάλλον από τη δική τους πλευρά στη δική μας. Πρέπει λοιπόν να ε, μπουν όλα αυτά στην έκθεση. Και επιπλέον θα ήθελα να πω ότι οι κύριες ανησυχίες των ε, Ευρωπαίων διπλωματών εκείνη την ε, περίοδο ήταν εάν οι κυβερνήσεις της Ένωσης θα δώσουν πραγματικά αυτά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και πώς θα τα δώσουν, με τι τρόπο θα ε, φτάσουν τα κονδύλια στην Τουρκία. Αυτό απασχολούσε και εμάς. Το ποιο δηλαδή θα διαχειριστεί αυτά τα κονδύλια όταν φτάσουν. Φυσικά πρέπει, θεωρώ, τα κονδύλια να διατεθούν μέσω της κυβέρνησης, μέσω των Υπουργείων, αλλά πρέπει να φτάσουν και στα σωστά χέρια. Αυτό που είδαμε επίσης είναι ότι υπάρχουν πάρα, πολλοί, πάρα πολλές ΜΚΟ που φροντίζουν για τη σύντηση ε, όμως υπάρχουν ελλείψεις οικονομικές, υπάρχει ελλείψη σε οργάνωση. Δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρετε, να ταΐσεις κόσμο που βρίσκεται και στο δρόμο. Και δεν μιλώ μόνο για τις ε, πόλεις. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένες ε, πόλεις που λένε ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας Τούρκος εδώ, όλοι Σύριοι είναι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να λάβουμε υπόψη την άποψη των ε, ΜΚΟ. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους τους και όλοι μας εξέφρασαν ανησυχίες για το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση στην Τουρκία. Διότι η κατάσταση χειροτερεύει. Μας είπαν ότι υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι Τούρκοι στην Τουρκία. Υπάρχει πρόβλημα με τους Κούρδους Γι' αυτό Εξαιτία τη εισρωή των προσφύγων, οι Κούρδοι και οι Τούρκοι φεύγουν από τα χωριά του. Επίση, δεν υπάρχει κανένα σεβασμό στι ε, ε, μειονότητε, καμία απολύτω ελευθεροτυπία. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλα προβλήματα ε, και πολιτική αστάθεια. Τώρα, ποιος τη χαρακτηρίζει σταθερή τη χώρα, ποιο όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όμως προσφυγική και μεταναστευτική κρίση έχει κάνει τα πράγματα ακόμα δυσκολότερα στην Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ. Η Ναταλή Κρίσπακ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Σιλβία Μαρία και η Τάνια άριστα υπενθύμησαν ε, τα διάφορα βασικά στοιχεία της αποστολής. Η αποστολή ήταν άκρως ενδιαφέρουσα, μας επέτρεψε σε ελάχιστες ώρες να λάβουμε γνώση των σημαντικοτάτων προβλημάτων σε αυτό το σημείο του κόσμου και μας υπενθύμησε πόσο μας προβληματίζει και μας αφορά τους Ευρωπαίους. Άκρος ενδιαφέρουσα ήταν η επίσκεψή μας, στα σύνορα με τη Συρία, στην περιοχή εκείνη που πλήττεται περισσότερο στην Τουρκία, όπως τον Καζεντέπ και στον καταβλισμό του Ιζίπ γινόταν διαπραγματεύσεις για την περίφημη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενώσεως Τουρκίας. Ε, το ποσό που ετίθετο τότε ήταν τρία δις, χάρη στην έξοχη διοργάνωση, για την οποία ευχαριστώ την Κατρίνη Μπέρ, τον Νικολά, τον Τόμ, την Ευαγγελία και τον Λιγκό για την υπομονή που μας έδειξαν διότι η Άννα Μαρία καμιά φορά έμενε πίσω και έπρεπε να την μαζεύουμε και να ξαναμπαίνει στο κοπάδι ε, ήταν λοιπόν πάρα πολύ καλά οργανωμένη η επίσκεψη όσον αφορά τη συναντήση με τις ΜΚΟ και με την ε, Συριακή Διασπορά που συναντήσαμε σε όλη τη την ποικιλομορφία και με τους διάφορους φορείς, τους αξιωματούχους συναντήσαμε. Τα πρακτικά το σημειώνουν αυτό άριστα, δύο τις παρατηρήσεις ε, έχω, διότι συμμερίζομαι απόλυτα τα υποθέντα όσον αφορά ε, ε, ε, πώς φροντίζανε τους πρόσφυγες. Ήταν πολύ ποιοτική η υποδοχή τους και η οργάνωση. Στη Γαλλία δεν είναι εξίσου καλή όσο η υποδοχή που γίνεται στην Τουρκία. Μία παρατήρηση. Στο Κίλης εδώ και 4,5 χρόνια είχα πάει και μετά από 4,5 χρόνια που πήγα στον καταβλισμό είδα πόσο η διπλωματική και η πολιτική θέση της μεγάλης αυτής χώρας που είναι η Τουρκία ε, είχε αλλάξει. Εδώ και 4,5 χρόνια ε, είχαν υποδεχτεί ήδη πάρα πολλούς ε, Σύρους που ξέφευγαν από τις βιοπραγίες και τον πόλεμο και πήγαν στην Τουρκία. Οι Τούρκοι θεωρούσαν την υποδοχή αδελφών και δεν ζητούσαν τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε. Άλλαξε όμως η κατάσταση. Ε, διότι μετά γίνηκαν οι διαπραγματεύσεις, συσχετίστηκα, συζητήθηκε η υποδοχή με την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα άλλη τοποθέτηση. Και δεν συνδεόταν μόνο με τον αυξανόμενο αριθμό των προσφύγων που καταφεύγουν στην Τουρκία. Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η βοήθεια ευρωπαϊκή θα πρέπει να έχει σαν στόχο την, την τοπική διάσταση να πηγαίνουν τα χρήματα όσο πιο κοντά στους πρόσφυγες γίνεται. Να επενθυμίσω λοιπόν ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις εντυπώσεις από την αποστολή που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες στα σύνομη της τη Συρία και να πούμε ότι τα προβλήματα είναι και δικά μας προβλήματα. Είναι τεράστια προβλήματα παρά μόνο με κινητοποίηση των κρατών μελών και με κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που όπως διαπιστώσαμε είναι τεράστια. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, γνωρίζετε, αυτές οι εκθέσεις πηγαίνουν στη διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών και στον Πρόεδρο Σούλτς. Όμως, ε, να σας πω ότι παρακολουθούσα ε, τις δραστηριότητές σας και στο Twitter και με μεγάλο ενδιαφέρον. και πιστεύω πως ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε για την οργάνωση και έμαθα πάρα πολλά από τις ε, ανταποκρίσεις σας. Πιστεύω πως μας εκπροσωπήσατε άριστα στον ε, λίγο διαθέσιμο χρόνο που είχατε. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη η βοήθειά σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε όλοι πόσο μεγάλη ε, και χρήσιμη δουλειά είναι αυτή που γίνεται από την Γραμματεία για την όλη διοργάνωση αυτών των αποστολών. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε με ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό σημείο στη Μεσή Διάταξη. Μιλώ για το σημείο 8 την ανακοίνωση της Επιτροπής ε, προς το Κοινοβούλιο του Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και προώθηση των νόμιμων οδών προς την Ευρώπη. Είναι μια παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρω... την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Άσυλο, την ΕΑΣΟ εστιάσαμε σε ε, δύο θέματα. Ε, εστίασε σε δύο θέματα η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τη μία προτείνονται μεταρρυθμίσεις για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για το άσυλο, ιδιαίτερα ε, αναθεώρηση του Δουβλίνου. Από την άλλη προτείνονται διάφορα μέτρα που θα ενισχύσουν την νόμιμη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την μπλε κάρτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα θα μας παρουσιάσει τις προτάσεις έτσι ώστε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Καταρχάς, η συζήτηση θα εστιαστεί στο πώς μπορεί να βελτιωθεί το κοινό σύστημα για το άσυλο, ιδιαίτερα από την πτυχή της αλληλεγγύης και ε, του καταμερισμού ε, εργασιών. Γι' αυτό θα ε, καλωσορίσουμε τον Τζον Πιερι Σκέμπρι από την ΕΑΣΟ, και στο δεύτερο γύρο των συζητήσεων θα εστιάσουμε στις νόμιμες οδούς προς την Ευρώπη. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Νίλσεν. Και πρώτα θα δώσουμε το λόγο σε εκείνον για να μας παρουσιάσει τις διάφορες επιλογές ε, που υπάρχουν για τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος για το άσυλο και μετά θα περάσουμε στον κύριο Σέμπρι. Στη συνέχεια θα λάβουν το λόγο οι ε, εισηγητές και οι σκιώδες εισηγητές για τις βασικές σχετικές εκθέσεις. Συνοψίζονταν λοιπόν, ο κύριος Νίλσεν και ο κύριος Έμπρη θα λάβουν πρώτοι το λόγο και μετά όλα τα μέλη της Επιτροπής και όλοι οι ε, εισηγητές βασικών σχετικών εκθέσεων. Κύριε Νίλσεν, έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ επίσης να είστε όλοι σύντομοι, διότι υπάρχει ε, λίγος χρόνος και είστε πολλοί όσοι θέλετε να λάβετε το λόγο. Έξι λεπτά περίπου έχετε, έξι-εφτά λεπτά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω αυτήν την πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος όπως μου ζητήσατε. Επί το παρόντος θέλουμε να εστιάσουμε σε βραχυπρόθεσμη εφαρμογή των ε, μέτρων ε, αντιμετώπισης της κρίσης. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό ε, να δούμε πως έχουμε εντοπίσει διαρθρωτικές αδυναμίες σε όλο το πλαίσιο του κοινού συστήματος για το άσυλο και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία και αναθεώρηση του όλου του πλαισίου μέσω και μακροπρόθεσμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε σωστά όλες τις ε, πιθανότητες ε, εισόδου προσφυγικών νερών στην Ευρώπη. Πρέπει να προσπατεύσουμε του ετούντε άσυλο και να διατηρήσουμε καταρχά δίκαιη και ίση μεταχείριση και μέσα στα κρατημέλη και προ του πρόσφυγες πρέπει να παρέχουμε νόμιμες ε, οδούς εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα αποθαρρύνει την παράτυπη εισρωή μεταναστών και προσφυγών στην Ευρώπη και έπειτα να γίνονται απόλυτα σεβαστά τα δικαιώματα των ε, προσφύγων και των ετούτων άσυλο. Καταρχά, προσπαθήσαμε να αναθεωρήσουμε όλα τα κύρια στοιχεία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματο για το άσυλο, όπω είναι σήμερα. Εντοπίσαμε ουσιαστικά πέντε προτεραιότητε και επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή νέε προτάσει. Καταρχά, αναθεώρηση του συστήματο του Δουβλίνου. Δεύτερον, έγκριση τη βάση δεδομένων τη Eurodac και τα δεκτυλικά αποτυπώματα. Τρίτον, σύγκληση προ την ίση μεταχείριση από τα κράτη-μέλη σχετικά με το ποιο αποφασίζει τι για τις ε, αιτήσει ασύλου. Τέταρτον, ε, ύπαρξη ενό καλύτερου πλαισίου για τις ε, δευτερογενείς μετακίνησει των ετούντων άσυλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος πώς θα ενισχύσουμε την ΕΑΣΟ. Πολύ σύντομα, καταρχάς ε, σχετικά με το Δουβλίνο, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει μια βιώσιμη ίση κατανομή ευθύνη σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έπειτα, πρέπει να επαναξετάσουμε το αν μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα ίδια κριτήρια για την παράτηση τύπη είσοδο σε ένα κρατό μέλο, και αν αυτό το κράτο πρέπει να είναι υπεύθυνο για την περαιτέρω επεξεργασία του αιτήματο ασύλου. Ε, έπειτα πρέπει να δούμε πώς θα επανασχεδιάσουμε το Δουβλίνο έτσι ώστε να περιοριστούν οι δευτερογενείς μετακινήσεις. Έχουμε δει ότι υπήρχαν ε, δευτερογενείς μετακινήσεις μεγάλης κλίμακας το 2015 και εδώ έχουμε εντοπίσει και διαρθρωτικά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα δεν θα ξεπεραστούν μόνο χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους κανόνες. Χρειάζονται... Ε, νέες προτάσεις που θα συμπληρώσουν το φυστάμενο πλαίσιο. Έχουμε εντοπίσει εδώ δύο επιλογές που ε, πρέπει να συζητηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρωτού αποφασίσουμε. Πρώτη επιλογή να διατηρήσουμε τα βασικά κριτήρια ε, που έχουμε όσο τώρα, δηλαδή ευθύνη του κράτους ε, μέλους πρώτης εισόδου και να ε, συμπληρώσουμε το σύστημα με έναν μηχανισμό ε, ίσης δίκαιης συμπεριφοράς μάλλον, που θα διευκολύνει την ανταλλαγή ε, πληροφοριών και θα ε, διευκολύνει επίσης την κατανομή του εφόρτου εργασία. Κάτι παρόμοιο μα παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι. Έπειτα, η δεύτερη επιλογή είναι μια πιο έντονη αλλαγή. Θα αλλάξει η ευθύνη από το κράτος μέλος της πρώτης εισόδου και έτσι όταν φτάνει κάποιος άνθρωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από εκεί θα ε, ε, χρησιμοποιείται ένα σύστημα αναδιανομής έτσι ώστε να υπάρχει ε, δίκαιη κατανομή. Χρειάζεται όμως θεμελιώδης αναδιάρθρωση του συστήματος. Επίσης, από αυτές τις δύο επιλογές μπορούν να δημιουργηθούν άπειρες υποεπιλογές. Το βασικό θέμα όμως είναι ζήτημα αρχής και εδώ θα θέλαμε τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να μας ε, πείτε τι πιστεύετε εσείς πως είναι ένα σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι έτσι θα έχουμε έναν επικοδομητικό ε, διάλογο. Τώρα, προτεραιότητες. Eurodac πρέπει να προσαρμοστεί ε, στις αλλαγές που θα γίνουν στο Δουβλίνο, έτσι ώστε να μπορέσουν να αλληλοσυμπληρώνονται. Έπειτα πρέπει να δούμε πώς θα επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή της ε, Eurodac για να καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση και να διευκολύνει την πολιτική επιστροφών. Έπειτα, σύγκληση και ε, πρόληψη δευτερογενών μετακινήσεων. Υπάρχει ένα ε, σχέδιο σχετικά με τις ε, συνθήκες υποδοχής και κράτησης. Έχουμε εντοπίσει αρκετά προβλήματα, παρότι οι οδηγίες είναι σχετικά πρόσφατες. Υπάρχει χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης στα κράτη-μέλη, υπάρχουν διαφορετικά καθεστώτα που ε, λαμβάνουν οι αιτούντες σε άσυλο, υπάρχουν διαφορετικά χρονικά διαστήματα που διαρκεί η επεξεργασία ενός αιτήματο σε... Με λίγα λόγια, αυτό που προσπαθούμε είναι να επιτύχουμε μία εναρμόνιση του συστήματος ασύλου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε οι οδηγίες να γίνουν κανονισμοί και να διευκολύνουν την ε, ομοιόμορφη και ίση εφαρμογή ε, των ε, νόμων. Τέλος, ο συνάδελφος από την ΕΑΣΟ θα σας μιλήσει για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την υπηρεσία σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Να σας πω επίσης ότι εργαζόμαστε πυρετοδό σε ένα πολύ ε, μικρό χρονοδιάγραμμα και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και τώρα στον κύριο Σαμπρί να παρουσιάσει τις απόψεις του φορέα που προσωπεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ λέει ο κύριος Κέμπρη Ευχαριστώ που καλείτε τον φορέα μας ε, να συμμετάσχει στη συζήτηση. Ο διευθυντής μας δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Ε, όμως μου ζήτησε να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του, ε, να σας συστηθώ. Είμαι υπεύθυνο για τις σχέσεις με τους ενδιαφερομένους φορείς και την επικοινωνία και θέλω να εκφράσω τις απόψεις μας σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οποία θα ακούσατε πολλά. Καταρχάς, ποιο είναι το γενικό πλαίσιο. Θα γνωρίζετε ότι έχουμε μεγάλη κλίμακα, αφήξει σε υψηλή κλίμακα και ε, μεγάλη κλίμακα και αυτό πιέζει τα κράτη-μέλη και το σύστημα ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 28 Ιουλίου του 2015 καταλήξαμε σε μια προθεσμία για την ενσωμάτωση εθνικό δίκαιο ε, των μέτρων αυτών. Πλησιάζει η πρώτη επέτειος. Η ΕΑΣΟ λοιπόν θεωρείται πλέον σημαντικός φορέας όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων και της παρούσης καταστάσεως. Αρκεί να πω ότι σήμερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας μάλιστα θα έχουμε 250 αξιωματούχους που θα ασχολούνται με το θέμα της υλοποίησης της συμφωνίας ε, ε, των, ε, της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ενώσης Τουρκίας σε Ελλάδα και Τουρκία. Πολύ ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς ποιο ήταν το δυναμικό μας πριν από μερικές εβδομάδες. Η παρούσα κατάσταση ποια είναι όσον αφορά το άσυλο. Υπάρχει νέος ρυθμός στην ΕΑΣΟ και επεκτείνεται ο φορέας μας. Άρα τώρα είναι σωστή στιγμή για να επανεξετάσουμε την εντολή που έχει δοθεί στον οργανισμό. Ε, σε αυτό το πλαίσιο καλωσορίζω την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την εντολή μας. Το σημαντικό εδώ είναι η εντολή να ταιριάζει καλύτερα στην αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε τώρα. Τι θα θέλαμε να δούμε στην εντολή. Θέλουμε να δούμε τέσσερα βασικά στοιχεία. Το πρώτο, ένα ρόλο όσον αφορά την εποπτεία των εργασιών μας και να έχουμε επιχειρησιακή δυνατότητα να κινηθούμε όπου αυτό απαιτείται. Τρίτον, να μπορούμε να εξασφαλίζουμε εναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας και τέταρτον, να παίξουμε ένα ρόλο στην, προτινό, στην εφαρμογή της προτινόμενης κλίδας κατανομής ε, του Δουβλίνου. Λοιπόν, καταρχάς, εποπτεία του ΣΕΑΣ. Σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην κρίση πιστεύουν ότι η μόνη αξιοπιστή λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Κανένα κράτος μέλος μόνο του μπορεί να λύσει το πρόβλημα της μετανάστευσης και της μεταναστευτικές ροές. Εναρμόνιση της νομοθεσίας είναι σημαντική. Αυτό όμως πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, των συμφωνηθέντων. Στην ΕΑΖΟ έχουμε ετοιμάσει πολλά εργαλεία, εκθέσεις, κατάρτιση προσωπικού σε όλο το φάσμα που καλύπτεται. Έχουμε δημιουργήσει επαφές με τα κράτη-μέλη και έχει δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ ημών και των ε, κρατών μελών και των άλλων εμπλεκομένων φορέων. Άρα τώρα μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα, δηλαδή να υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος ομοιόμορφης εφαρμογής της ε, θεσπιστής νομοθεσίας. Το δεύτερο, αφορά τα επιχειρησιακά, το επιχειρησιακό δυναμικό του οργανισμού. Πρέπει να μπορούμε να παρέχουμε κατεπηγόντως βοήθεια όταν αυτή απαιτείται. Πρέπει να δρομολογούνται τα δέοντα μέτρα. Η κρίση έδειξε ότι σαν οργανισμός ασύλου πρέπει να μπορούμε να ανατήσουμε το δυναμικό μας, το προσωπικό μας τάχιστα. Για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε προσωπικό προφανώς. Ανθρώπους. Και να έχουμε ε, και δυνατότητα συμπληρωματικού προσωπικού. Ε, χρειαζόμαστε τους δικούς μας, τη δική μας ομάδα τόσο το ΕΑΣΟ, που μαζί με τη βοήθεια που θα παράσχεται από τα κράτη-μέλη να μπορούμε γρήγορα να αναπτύσσουμε το δυναμικό, το προσωπικό μας στην περιοχή όπου αντιμετωπίζεται κρίση. Τρίτον, πρέπει να εξασφαλίσουμε εναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας εναρμονισμένη νομοθεσία σχετίζεται με συνεκτική και πλήρη εφαρμογή αυτής. Εδώ εκδίδουμε εκθέσεις όσον αφορά τις χώρες καταγωγής, αλλά δίνουμε και τεχνογνωσία μας για να αναλύουμε όλα τα σχετικά ε, κείμενα που αφορούν και την κατάσταση τρίτες χώρες. Έτσι τελικά οδηγούμεθα σε ομοιόμορφη εφαρμογή όπως, αρχών όπως είναι η ασφαλής χώρα καταγωγής, ασφαλής ε, τρίτη χώρα και ασφαλής χώρα χορηγήσεως ασύλου. Πρέπει να εφαρμόζουμε σωστά τα απορίσματα των εκθέσεων. Και έτσι να λαμβάνονται και αποφάσει για τη χορήγηση ασύλου με πιο μειομορφό τρόπο. Και έχουμε και πρόγραμμα κατάρτισης. Πάνω από 10.000 ανθρώπου έχουμε εκπαιδεύσει. Αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε περισσότερου. Πιστεύουμε ότι αν πάμε στο ίδιο σχολείο καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα. Αυτό που θα θέλαμε λοιπόν θα ήταν κάποια από τα μαθήματα να γίνονται υποχρεωτικά. Να διδάσκονται στα κράτη-μέλη τους ώστε να εκπαιδεύονται περισσότερο, ε, περισσότεροι άνθρωποι και να κάνουν τα ίδια μαθήματα. Το τέταρτο κομμάτι αφορά την κλίδα κατανομής του Δουβλίνου. Εδώ σημειώνουμε τον αξανόμενο ρόλο. που αναφέρεται στην, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το φορέα μας. Έχουμε την εμπειρία σαν ΕΑΖΟ όσον αφορά τις μετεγκαταστάσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα και την Ιταλία. Και θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Η κλίδα ε, βασίζεται σε σαφή κριτήρια. Αυτό θα διευκολύνει την εφαρμογή, αν υπάρχουν σαφή κριτήρια. Και έτσι τελικά θα υπάρχει κοινή αντιμετώπιση των ευθυνών και θα επικρατήσει αλληλεγγύη. Αν κατακλείδη. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να τονίσω και το εξή. Οι συμπληρωματικοί ρόλοι που μας ανατίθενται ή που θα μας ανατεθούν, ελπίζουμε, θα σημαίνει ότι θα χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, χρήματα και ανθρώπους. Ε, εκατό περίπου άνθρωποι δεν μπορούν να πετύχουν όλους τους στόχους και να ανταποκριθούν στα καθήκοντα. Θα χρειαστούμε λοιπόν επαρκείς ανθρωπίνους πόρους, προσωπικό. Και το Κοινοβούλιο επανειλημμένα ζήτησε κάτι τέτοιο. Περισσότερους πόρους για το ΕΑΖΟ Κάτι που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στο ψήφισμά σα τη 12η Απριλίου που αφορούσε την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη ολιστική προσεγγίσεω. Κάτι που καλωσορίζουμε και σα ευχαριστούμε γι' αυτό. Συνάδελφοι, έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Σέμπρη και τον κύριο Νίλσεν. Έχουμε ένα θεματάκι εδώ. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να ασχοληθούμε με ένα τόσο πολύπλοκο θέμα. Έχουμε την έκθεση για τους ξένους μαχητές που είναι προγραμματισμένη να εξεταστεί στις 11.30 και μπορεί να αργήσουμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μέλη που θέλουν να ε, είναι παρόντα εκεί. Έχω 13-14 μέλη της Επιτροπής που ζήτησαν το λόγο και η συζήτηση θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το δεύτερο μέρος ε, θα ε, είναι σχετικά με την ε, νόμιμη μετανάστευση. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από όλους όσους, όλους όσοι θέλετε το λόγο, τους εισηγητές και σχεδόν εισηγητές σχετικά με το Δουβλίνο και όλα τα άλλα σχετικά θέματα, να ε, αναφερθείτε στην ανακοίνωση έτσι όπως ε, την έχετε διαβάσει. Διαφορετικά δεν θα προλάβουμε χρονικά. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο περίπλοκο θέμα και θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω τα σχόλιά σας για την ανακοίνωση. Όπως σας είπα, 14 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Προσπαθήστε λοιπόν να ε, μιλήσετε το πολύ δύο λεπτά κύριος ε, Λέναρτ έχει το λόγο. Θα δώσω το λόγο σύμφωνα με τη σειρά, με τη σειρά που ε, ζητήθηκε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρουσιάσεις. Πιστεύω πως θα ήταν καλό να κοιτάξουμε και τη μακροπρόθεσμη προοπτική εδώ και όχι μόνο τον ε, μηχανισμό ε, άμεσης επίλυσης κρίσεως, κρίσεων. Μου έκανε εντύπωση η πρώτη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι μου φαίνεται πως υπάρχει έλλειψη ανατολισμού. Αναρωτιέμαι, και τα δύο συστήματα που μας παρουσιάστηκαν και οι δύο επιλογές μπορούν να λειτουργήσουν σωστά μόνο όταν και τα 28 κράτη-μέλη ε, είναι πρόθυμα να τις εφαρμόσουν στην πράξη. Είδαμε με τους μηχανισμούς κατάσταση στην περίπτωση της Ελλάδας και της Ιταλίας ότι η προθυμία των κρατών μελών ε, δεν υπάρχει. Θα μπορούσε λοιπόν μακροπρόθεσμα να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σχέδιο. Ε, Αυτά ως προς το μακροπρόθεσμο σκέλος. Τώρα, πρόθεσμα οι δευτερογενής μετακινήσεις, η ε, διεύρυνση του, ε, της χρήσης του συστήματος Eurodac. Εδώ πιστεύω πως ε, θα μπορούσαμε να δράσουμε πολύ πιο γρήγορα και δεν χρειάζεται να περιμένουμε την παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι γρήγορη, να παρουσιάσει τις προτάσεις σύντομα για να μην χρειαστεί να περιμένουμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Ε, πράγματι, ε, έχετε δίκιο. Η κυρία Βίξτρομ τώρα έχει το λόγο που ήταν η εισηγήτρια για τον ε, κανονισμό του Δουβλίνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ναι, γενικά θα πω ότι θεωρώ την έκθεση αρκετά καλή. Είναι κάτι που μας εμπνέει, δείχνει ηγετικέ ικανότητες, ε, μάλιστα σε μια εποχή όπου με ελάχιστες εξαιρέξεις οι Ευρωπαίοι ηγέτες ε, είναι απόντες από την ε, όλη συζήτηση. Θέλω να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει την έγκριση που έγινε τελευταία εβδομάδα στο Στρασβούργο για την ε, ολιστική προσέγγιση στη μετανάστευση. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δύο ψηφίσματα τα οποία ε, εγκρίθηκαν πέρυσι, όπου ήταν σαφέστατο το πολιτικό μήνυμα. Ήταν σαφέστατη η κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να προχωρήσουμε και είχαμε τεράστια στήριξη. Τι έχει συμβεί εδώ. Έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα ίσης κατανομής του φόρτου εργασίας και σχετικά με τις ε, αιτήσει ασύλου. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ότι μόνο ελάχιστα από τα 28 κράτη-μέλη έχουν συνεισφέρει πραγματικά ε, στην προσπάθεια αυτή. Επίσης, ε, σύμφωνα με την επιλογή Δύο της ε, ανακοίνωσης ε, πρέπει να υιοθετήσουμε μια ολιστική προσέγγιση στην μετανάστευση. Και σε αυτό με βρίσκεται σύμφωνη. Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνήσει σε αυτό θα βρει μεγάλη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορώ να προβλέψω Μάλλον δεν μπορώ, να, μαντέ, δεν μπορώ να, να φανταστώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να δεχτεί οτιδήποτε λιγότερο από αυτά που προτείνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιώμη έχει το λόγο που είχε αναλάβει την έκθεση για τις ασφαλείς χώρες ε, καταγωγής. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται όσον αφορά τον κανονισμό του Δουβλίνου και την κλίδα κατανομής ε, που πρέπει για το η είναι σωστό. αυτά είναι παλιά πορίσματα. Η παρούσα κρίση κατέδειξε ότι οι αρχές λειτουργίας πρέπει να αλλάξουν το συστημάτων. Αν ο κανονισμός του Διβλίνου πρέπει να τροποποιηθεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο αν παράλληλα οι, διαδικ... οι συνθήκες υποδοχής ε, στα κράτη-μέλη εναρμονιστούν. Αυτό που βρίσκω αρκετά ανησυχητικό στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δημιουργείται η εντύπωση ότι μόνο οι διατάξεις οι πιο περιοριστικές στοχεύονται. Οι κυρώσεις ε, ε, όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και νομίζω ότι πολλά στην ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται και δεν γίνεται σωστός υπολογισμός. Σε αυτή τη φάση δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να βασιστούμε σε θετική εξέλιξη και λειτουργία του συστήματος για την κατανομή ε, των ετούντων άσυλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα πρέπει να είναι πιο επιτυχές. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι επιτυχές το σύστημα. Πώς μπορούμε να βασιστούμε σε σωστή κατανομή και αν υπάρξει πρόοδος στα κράτη-μέλη θα είναι ε, περισσότερο, θα βασίζεται στη βούληση παρά στο σύστημα. Θλιβερή ηρωνία της ιστορίας. Πρόσφατα μάχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει πιο φιλόδοξο κανονισμός του ασύλου. Κάπου κολλάει, βέβαια, στα κράτη-μέλη και αυτή η προσπάθεια κολλάει σε, ε, σε ένα μποϊκοτάζ από την αρχή που γίνονται τα κράτη-μέλη. Κολλάει στα τείχη των κρατών μελών. Ζητάτε την άποψή μας. Στα πρώτα στοιχεία της πρότασης. Υποστηρίζω το, την επιλογή 2 για τον κανονισμό του Διβλίνου. Σύστημα κατανομής βάση κλίδας. Ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται σύστημα αποζημιώσεων, αντισταθμίσεων. Μακροπρόθεσμα θα δοθεί σε μια σούπερ εάζο μεγαλύτερη ευθύνη. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και εδώ τίθεται και το θέμα της εντολής που θα δοθεί στο ΕΑΖΟ. Τι άλλο παρατηρώ. Να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τροποποίηση των άλλων κειμένων για το κοινό καθεστώς ασύλου. Οδηγία περί διαδικασιών, οδηγία περί προσόντων και οδηγία περί υποδοχής. Μπορούμε να βρούμε λύση μέσω κανονισμών για να πετύχουμε σύγκληση όσον αφορά την αίτηση ασύλου. Χρειάζεται επαγρύπνηση. Όσον δεν θέλουμε να αποκτήσουν οι αλλαγές χαρακτήρα ποινών που επιβάλλονται. Με απογοητεύουν οι προτάσεις που γίνονται όσον αφορά την νόμιμη μετανάστευση. Δεν υπάρχουν πολλά καινούργια στοιχεία σε αυτά που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματικό θα είναι το σύστημα μεταεγκατάστασης. Αυτά είναι τα σχόλια που είχα. Um, Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Η Κορνιλία. Ευχαριστώ, Κλοντ. Έχω τρία πράγματα να πω. Πρώτο, κάτι ε, που είπαν και άλλοι συναδελφοί μου πριν. Έχουμε δηλαδή μια, ένα, ένα μηχανισμό ε, αντιμετώπισης κατεπηγουσών καταστάσεων στα πλαίσια του Δουβλίνου. Δεν αρκεί. Αν μείνουμε εκεί, δεν χρειάζεται καν οποιαδήποτε μεταρρύθμιση τη συμφωνία του Δουβλίνου. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή καταστροφικό τρόπο. Δεύτερο, όντω χρειαζόμαστε μια κλίδα κατανομή. Η κλίδα κατανομή πάει να πει όμω, συνεπάγεται όμω, την ανατροπή του Δουβλίνου διότι το Δουβλίνο έχει μία βάση. Εκεί όπου φτάνει ο παράτυπος μετανάστης, εκεί ή ο πρόσφυγας, εκεί γίνεται η πρώτη καταγραφή και επεξεργασία της αίτησή του. Ούτως ή άλλως αυτό έχει αποτύχει. Τα λένε αυτά και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για Ιταλία και Ελλάδα. Άρα χρειαζόμαστε κλίδα κατανομής. Αυτό είναι σωστό. Στην ε, εν λόγω κατανομή πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και όλες τις διάφορες ε, διασυνδέσεις οικογενειακές και άλλες και στις περιπτώσεις των προσφύγων. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δηλαδή δεν έχει νόημα να στείλετε κάποιον στη Λιθουανία, ας πούμε, το λέω έτσι κάπως ομά, ας πούμε, ο οποίος έχει οικογένεια στη Γαλλία. Αυτά είναι ανοησίες. Το νόημα θα πρέπει να είναι, και αυτό μπορώ να το υποστηρίξω, ο άνθρωπος αυτός να φτάσει κάποια στιγμή στην οικογένειά του. Άρα πρέπει να δούμε τους οικογενειακούς δεσμούς, και να διατυπωθούν ξεκάθαρα κριτήρια. Νομίζω ότι αυτά είναι εφικτά. Για αυτή την δευτερεύουσα ας πούμε, μετανάστευση δεν πρέπει να την εξετάσουμε με τρόπο διακριτικό και επομένως ε, μειονεκτικό. Θα πρέπει ε, να μπορέσει το πρόσωπο να πάει να διαμείνει εκεί όπου έχει δεσμούς. Δεύτερο, Εάσω. Δεν μπορώ να φανταστώ οι μηχανισμοί λήψεως αποφάσεων να ανατίθεται στον οργανισμό αυτό. Για το άσυλο δηλαδή. Υπάρχει κάποια προστιθέμενη αξία, σύμφωνη, ότι κλείνουν δηλαδή κάποιες τρύπε για ε, τις διαδικασίες υποβολής ασύλου σε άλλες χώρες. αυτό ε, ε, εξαρτάται λίγο και από το επίπεδο. Είναι πλεονέκτημα υπέρ των προσφύγων. Εγώ δεν νομίζω, ούτε μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και με αύξηση του προσωπικού που ζητήσατε και για τον έλεγχο της εφαρμογής του συστήματος ασύλου, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, τι να σας πω τότε, καλή τύχη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτά μπορούν να κινηθούν μέσω του οργανισμού αυτού. Δεν εκφράζω κάποια δυσπιστία απέναντί σας, θεωρώ όμως ή τέλος πάντων διερωτώ με μήπως είναι παραπάνω από θα μπορείτε να κάνετε. Ευχαριστώ κύριε Σαρτζεντίνη. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι χρειάζεται μια σε βάθος μεταρρύθμιση. Πράγματι αυτό είναι το νόημα του κειμένου που έχουμε μπροστά μας. Συμφωνώ βέβαια με την ανάγκη εναρμόνισης του συστήματος ασύλου και μετανάστευσης. Οι οδηγίες να μετατραπούν σε κανονισμούς μου φαίνεται καλή ιδέα. Εξαρτάται βέβαια από το επίπεδο εναρμόνισης, από το επίπεδο ποιότητας, από το επίπεδο των δικαιωμάτων. Εάν εναρμονίσουμε στο επίπεδο του ε, του κοινού παρονομαστή, έχουμε πρόβλημα. Η ανακοίνωση λέει για παράδειγμα για την Qualification Directive λέει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και δευτερεύουσες μετακινήσεις. Εδώ μιλούμε για άσυλο και για πρόσφυγες. Και αν θέλουμε να εξετάσουμε τέτοιους παράγοντες μέσω της ε, ε, οδηγίας αυτής, νομίζω ότι πάμε πιο πολύ να μειώσουμε το επίπεδο των ε, ε δικαιωμάτων. Επίσης, ο έλεγχος για την ε, επικουρική προστασία. Σωστός έλεγχος. Αυτό σημαίνει όμως όσο περισσότεροι έλεγχοι ότι μπορεί να γίνει πιο εύκολη και πιο ταχεία η επικουρική προστασία. Σε ό,τι αφορά την οδηγία τώρα για τους όρου και τις συνθήκε υποδοχή. μα τα κάναμε αυτά πρόσφατα και τα εφαρμόζουν οι χώρε μέλη. Πάλι εκεί χρειάζεται εξασφάλιση ότι δεν θα γίνει κατάχρηση των δικαιωμάτων. Αλλά πάλι εκεί κατεβαίνουμε σε χαμηλότερο επίπεδο. Τώρα, κυρώσει για τι δευτερεύουσε μετακινήσεις για να μην καταχρώνται τα πρόσωπα αυτά των δυνατοτήτων αυτών. Είμαστε βέβαιες ότι μπορεί να γίνει αυτό. Πώς θα κριθεί ότι αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος είναι δευτερεύουσα κίνηση. Αυτά τα λέει η ανακοίνωση. Εγώ νομίζω μάλιστα ότι αυτό είναι παράνομο. Δηλαδή μια αίτηση ασύλου να πάει ως δευτερεύουσα μετακίνηση. Αυτό που μου φαίνεται ότι λείπει είναι οι νόμιμες οδοί εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμώ βέβαια το σχεδιασμό της ΆΣΟ, αλλά αυτό που λέει η ανακοίνωση κατά τη γνώμη μου, όπως τη διαβάζω εγώ, είναι ότι η χορήγηση περαιτέρω εξουσιών στην ΆΣΟ για να εναρμονίσει σε υψηλότερο επίπεδο τις πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης είναι περισσότερο μακροπρόθεσμα πράγματα. Αυτό ε, κατανοώ εγώ από την ε, ανακοίνωση και αυτό μου φαίνεται ότι δεν είναι υγιές. Άρα, με λίγα λόγια και ειλικρινώς, αν αυτή είναι η απάντησή μας στην κρίση του προσφυγικού, μου φαίνεται μια αναζήτηση νομοθετικών λύσεων, ώστε λιγότεροι να έρχονται τελικά εδώ και όχι να διευκολύνουμε ανθρώπου οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν από τον πόλεμο ή από τις δικτατορίες. Τέλος, χτες δεν μάθαμε, δεν έχουν αρκετό φαγητό τα μωρά στους προσφυγικούς καταβλημούς στην Ελλάδα. Κοιτάξτε κάποια σύντομα στοιχεία αν επιτρέπετε. Για το θέμα της ε, μετεγκατάστασης. Λοιπόν, κοιτάξτε πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση και το άσυλο ξεχωριστά, σαν ξεχωριστού τομεί. Τα δύο θέματα απαιτούν διαφορετικέ προσεγγίσεις. Δεύτερον, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μεγαλύτερη σύνδεση με την υπατή αρμοστία του ΟΗΕ για τα συστήματα μετεγκαταστάσεως. Αυτό πρέπει να γίνει ταχύτερο δυνατόν. Νομίζω ότι στις διαπραγματεύσεις μας με τρίτες χώρες όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες και το θέμα της ε, διανομής της ε, ξένης βοήθειας ε, χρειάζεται να το συζητήσουμε και να έχουμε συμφωνίες επανεισδοχής και να συνδεθούν μεταξύ τους. Για το Δουβλίνο νομίζω ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προσπαθεί να επανεφευρίσκει τον τροχό και υποστηρίζω την επιλογή για το Δουβλίνο που συντηρεί την αρχική αρχή να αιτείται το άσυλο στην πρώτη χώρα άφηξη και να έχουμε ένα σύστημα μετεγκατάσταση που θα βασίζεται και στις δικές μου προτάσεις ελπίζω. Φοβάμαι όταν δημιουργήσουμε ένα σύστημα όπου ουσιαστικά ζητά άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη και να ομαδοποιούνται τα αιτήματα ασύλου αυτό θα διατηρεί στα κράτη-μέλη εκείνα που τώρα έχουν μεγάλη πίεση πάνω τους μόνιμα τα στρατόπεδα διαμονής, ε, του ε, τους καταβλισμούς διαμονής. Χρειάζεται καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των βάσεων δεδομένων με τη σωστή προστασία αυτών. Αυτό θα μας βοηθούσε. Νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό να δούμε ε, την οριζόντια αναθεώρηση ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά το εμπόριο ανθρώπων και τη σύγχρονη ε, δουλεία. Υπάρχουν πολλά κενά, έχουμε πολλές διώξεις, αλλά δεν έχουμε αρκετές καταδίκες και επιβολή κυρώσεων. Και νομίζω, διότι υπάρχουν πολλά κενά και πρέπει να έχουμε σαφή πολιτική όσον αφορά την ένταξη στην κοινωνία και την συμπερίληψη των μεταναστών και των προσφύγων σε αυτές τις προσπάθειες. Εάν καλυπτόταν αυτές οι πτυχές, εγώ θα ήμουν πολύ πιο ικανοποιημένος με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, λέει η κυρία Μπιόρκ, κάποιες από τις ανησυχίε μου καλύφθηκαν τους συναδέλφους. Νομίζω ότι ναι το έγγραφο με τις προτάσεις του δίνει την εντύπωση πολλών κατασταλτικών ε, ε, μέτρων. Αναφέρεται σε παράγοντες ομαδοποίησεως ε, και κινούνται όλες οι προσπάθειες στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Οι νέοι κανονισμοί δεν ενθαρρύνουν τους πρόσφυγες να ζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη. Θέλουμε ευρωπαϊκές λύσεις. Αν βασίζονται επί αυξήσεως της ευθύνης για υποδοχή των προσφύγων. Αν αφορούν τα μέτρα για στατικοποίηση των συνόρων και να σταματήσει τον κόσμο το να έρχεται, αν αυτή είναι η προσέγγιση, είναι αδύνατο να στηρίξουμε τους κανόνες. Υπόθηκαν πράγματα για το Δουβλίνο. Πρέπει να πάμε στη δεύτερη επιλογή. Με κάποιες επιφυλάξεις βέβαια. Δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε προς στήριξη κανονισμών αν έχουν τη μορφή που έχουν στο έγγραφο. Να σταθώ στο θέμα της μετεγκαταστάσεως. Θα είμαι εισηγήτρια, βλέπετε, για το κοινοβούλιο από αυτού. Και πάνω σε αυτό, από ό,τι βλέπω στο έγγραφο, υπάρχει τάση να γίνεται, να συνδέεται με την κατάσταση με συμφωνίες με τρίτε χώρες. Έτσι στευλώνεται ένα μηχανισμό που βασίζεται επί διεθνού αλληλεγγύη και προστασίε ευαλώτων, προσφύγων που ζητούν ε, ασφάλεια στην Ευρώπη. Αν στευλωθεί ο μηχανισμό, διότι θα συναρτάται από συμφωνίες τωρινέ και μελλοντικέ, όπως αυτή με την Τουρκία που επικρίνουμε σαν κοινοβούλιο τότε αυτός δεν είναι σωστός δρόμος. Το λέω αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να μην προτείνουν τέτοιες λύσεις στις επικείμενες προτάσεις τους. Νομίζω ότι λείπει η αναφορά στους νόμιμους και ασφαλείς δρόμους, ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές. Δηλαδή το έγγραφο εμπεριέχει πολλά προβλήματα. Θα είσαι εισηγήτρια για την μετεγκατάσταση, πρέπει να το πω αυτό, ναι, ναι, το ξέχασα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μουσολίνη έχει το λόγο. Πρόεδρε, θα επικεντρωθώ επί της επιλογής 2, διότι επιλογή παριθμών 1 ε, δείχνει ότι έλλειψη βούλησης είναι απλώς ε, μια κοινή επιχείρηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι απέτυχε η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έστω και συμβολικά, έστω και τυπικά, να ενταχθεί σε όλες τις εδώ έχουμε ελάχιστη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρωταγωνιστούν τα κράτη-μέλη. Ε, τα λαμβάνω αυτά υπόψη. Βλέπω ότι έχει μεγάλο θάρρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα προτείνει. Να αποσυνδέσει τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ κράτους εισόδου, χώρας εισόδου και, και αιτήματος ασύλου. Αυτή η σύνδεση πρέπει να διακοπεί. Πώς. Όχι μόνο μέσω συμβαστικής λύσεως, δηλαδή μέσω της κλίδας κατανομής, που σίγουρα είναι καλή λύση, αλλά θέλουμε να δώσουμε στην ΕΑΣΟ επίσης περισσότερη δικαιοδοσία, μεγαλύτερη δικαιοδοσία. Η ΕΑΣΟ είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και κομμάτι των κρατών. Δεν είναι τεχνικός φορέας αποκλειστικά. Να δώσουμε και ψυχή στην ΕΑΣΟ. Δεν μπορούμε να πούμε δεν μπορεί να αξιολογεί και να αποφασίζει η ΕΑΣΟ μόνο μέσω μιας ανώτερης θέσεως θα τις δώσουμε, ανώτερη από τα κράτη-μέλη θα καταφέρουμε να αποφύγουμε τους εγωισμούς όλους αυτούς που υπάρχουν και να ενισχύσουμε και την Eurodac. Ενίσχυση τι σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Eurodac. Αυτό δεν ισχύει ακόμα. Εγώ ε, είδα ποια είναι τη συμφωνία του ΠΡΟΜ που υπεγράφει από την Αυστρία συμπτωματικά, την Αυστρία που σε αυτή τη φάση δημιουργεί τείχους, χαλάκι ε, στο Μπρένερ χτίζει. Παραβιάζει δηλαδή τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα πρέπει να υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία. Αυτό πρέπει να φανταστούμε. Η Ιταλία, το χάρη, τη συνθήκη του Προύμ το 2005 την παρέλαβε το 2009, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί ακόμα. Το, το στήριξε, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί ακόμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα κράτη-μέλη να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του Eurodac. Όχι μόνο να τα διαβιβάσουν, αλλά να έχουν και πρόσβαση. Άρα, ενίσχυση της ΕΑΖΟ και της Eurodac. Υπενθυμίζω ότι το Eurodac μπαίνει και στο νέο κανονισμό της Frontex και στην Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και τη μεθοριακή, ε, την Αρχή για Προστασία των Συνόρων και το έγγραφο περί παναπατρισμού και απελάσεως των παράτυπων μεταναστών. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και πολύ σημαντική είναι η διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων συστημάτων ελέγχου διότι ακόμα δεν υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Ξανά λέω, περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων οργανισμών για τα θέματα αυτά. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζήπαλη, αυτόν το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφέρθηκαν ήδη πάρα πολλά, γι' αυτό θα προσπαθήσω να εστιάσω σε ορισμένα στοιχεία αυτό. Ε, ο κύριος Νίλσεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι το 2015 απέδειξε ότι το σύστημα του Δουβλίνου δεν λειτουργεί. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Εδώ και χρόνια γνωρίζουμε ότι το Δουβλίνο δεν λειτουργεί. Και αρκετοί συνάδελφοι εδώ και εκτός Κοινοβουλίου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ζητούν κάτι νέο. Εγώ εκπλήσωμαι και ενοχλούμε μάλιστα κιόλας, διότι τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο φέτος, μετά από τόσον καιρό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους έκανε λόγο για μια αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου. Και τι έχουμε τώρα, για άλλη μια φορά, μια ανακοίνωση. Συγγνώμη, εγώ περίμενα ένα σχέδιο πρότασης για μια νέα οδηγία ή ένα νέο κανονισμό, όχι μια ανακοίνωση. Επίση, γίνεται λόγο για δευτερογενή μετακίνηση και για τρόπου ελέγχου. Δηλαδή τι εννοούμε, κάντε τι συνθήκε όσο το δυνατόν δυσκολότερε, έτσι ώστε να μην έρχεται κανεί. Ελπίζω όχι. Ελπίζω να μην εννοείται αυτό. Όταν ε, μιλάτε για δευτερογενή μετακίνηση, αυτό συμβαίνει καταρχάς για επανένωση με την οικογένεια και δεύτερον εξαιτίας έλλειψης πραγματικών πληροφοριών προς τους πρόσφυγες για τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν και τις ε, πιθανότητες, τις ρεαλιστικές πιθανότητες που έχουν να πάνε σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Αυτό θα ήθελα λοιπόν να γνωρίσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι ο κύριος Νίλσεν πολλές φορές έκανε λόγο για καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Τι εννοείται με αυτό. Κάθε μετανάστης Προ το παρόν, κάθε μετανάστης που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παράτυπος μετανάστης. Ακόμα και εκείνοι που φεύγουν από τη Συρία, από την Ερυθρέα, όλοι αυτοί είναι παράτυποι. Η καταπολέμηση λοιπόν της παράτυπης μετανάστευσης ναι. τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάθε φορά που θα χτυπάει την πόρτα μας ε, κάποιος και θα ζητά άσυλο θα του λέμε φύγε είσαι παράτυπος. Πώς επίσης θα χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια του ε, καταπιστεύματος για την Αφρική για να ε, βελτιώσουμε την ε, διαχείριση των συνόρων στην Σομαλία, το Σουδάν και την Ερυθρέα. Τι σημαίνει αυτό ως αποτέλεσμα, ότι εκείνοι που φεύγουν από τα βασανιστήρια θα αναγκαστούν να μείνουν εκεί. Αυτό σημαίνει δηλαδή καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Και αν όχι, τι σημαίνει. Τώρα, σχετικά με το σύστημα ασύλου, συμφωνώ απόλυτα ότι χρειάζεται περαιτέρω εναρμόνιση. Όχι όμως για να αποδυναμωθεί. Πρώτα πρέπει να δούμε εάν όλες οι οδηγίες και οι κανονισμοί έχουν διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται από όλα τα κράτη-μέλη. Και κάτι τελευταίο για την νόμιμη μετανάστευση. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τα πράγματα. Όταν μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση και αιτήματα ασύλου σημαίνει ανθρωπιστική βίζα, σημαίνει επανεγκατάσταση. Όταν μιλάμε επίσης για προστασία των ετούντων ασύλων δεν πρέπει να μιλάμε για προϋποθέσεις Η διαφορά, η διαφορά είναι ότι ορισμένοι ε, άνθρωποι φεύγουν από την ανέχεια και ψάχνουν μια καλύτερη ζωή και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτή είναι η διαφορά των, ε, του τον από τους μετανάστες. Πρέπει να βρούμε διάφορους τρόπους να επεκτείνουμε για παράδειγμα την μπλε κάρτα, αλλά χρειάζεται προσοχή όταν συζητάμε και όταν προσπαθούμε να τα ε, συμπεριλάβουμε όλα σε ένα έγγραφο, διότι δεν πρέπει να συγχέονται ε, αυτά τα θέματα. Η κυρία Χολμάιρ έχει το λόγο. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό που μας παρουσίασε. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση την οποία πρέπει να δούμε ρεαλιστικά. Πρέπει να έχουμε οράματα, πρέπει να έχουμε επιθυμίες, όμως τα κράτη-μέλη πρέπει καταρχάς να συμφωνήσουν, δεύτερον να εφαρμόσουν και ε, τρίτον να έχουν τις δυνατότητες να ε, εφαρμόσουν αυτές ε, τις... Αυτό πρέπει να εφαρμόσουν. Η από την άλλη, έχω να πω ότι όταν η ΕΚΟΥ έχει μέλη που είναι κυβέρνηση στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνα για το ότι δεν έχουν να φάνε τα μωρά που φτάνουν ε, ως πρόσφυγες, τότε υπάρχουν ευθύνες. Φυσικά και είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι στην Ελλάδα περιμένουν ώρες στην ουρά οι άνθρωποι για να πάρουν κάτι να φάνε και όταν έχουμε 50.000 πρόσφυγες ε, θα έπρεπε ε, να είναι σε θέση η κυβέρνηση στην Ελλάδα να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Και... Ε, και η ΕΑΣΟ και η Frontex και διεθνείς οργανισμοί έχουν προσφέρει βοήθεια και έχει ε, παρατηρηθεί μεγάλη καθυστέρηση μέχρι να δεχτεί η ελληνική κυβέρνηση τη βοήθεια και να την χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ε, αναφέρουμε, πρέπει να αναφέρουμε τα πράγματα όπως είναι και να το ε, εξετάσουμε. Επίσης, ΕΑΣΟ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε περίοδο κρίσης όμως πιστεύω ότι το πακέτο για το άσυλο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο για να ε, διασφαλιστεί ε, η σωστή ε, ποιότητα στην ανταλλαγή πληροφοριών έτσι ώστε όλα τα κάτι μέλη να μπορούν να συνεισφέρουν. Χρειάζεται φυσικά και αναδιάρθρωση της ΕΑΣΟ έτσι να μπορέσει να αναλάβει και να εκτελέσει τα καθήκοντά της και τα νέα καθήκοντα που θα της ανατεθούν και αυτό ε, χρειάζεται την ευρεία στήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που δεν ε, συμβαίνει πάντα. Ε, γι' αυτό εμεί πρέπει να στηρίξουμε την ΕΑΣΟ, διότι πολλέ φορέ δεν βρίσκεται στήριξη από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να τη δώσουμε την νομιμότητα έτσι ώστε να μπορέσει να εκτελέσει τα καθήκοντά τη. Επίσης, θα ήθελα να στηρίξω την άποψη του Τίμωθη Κέρκο, ο οποίος ε, μίλησε για την επανεγκατάσταση. Πράγματι, χρειάζεται επίσπευση των διαδικασιών επανεγκατάστασης. Πιο γρήγορες αποφάσεις, πιο γρήγορες αποφάσεις και από την Ιντεπατή για τους πρόσφυγες και από τους ε, διεθνείς οργανισμούς. Όταν μια τέτοια απόφαση κρατά μέχρι 10 ε, μήνες, τότε δεν δίνεται κανένα κίνητρο ε, για να ζητήσουν οι ίδιοι άνθρωποι να επανακατασταθούν κάπου αλλού. Επίσης, ε, πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους για υποδοχή προσφύγων και όχι μόνο με μονομένα άτομα, αλλά όλες τις οικογένειές τους, έτσι ώστε να μπορέσουν οι οικογένειες να επανενωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αισθάνονται ότι δεν σκορπίστηκαν. Τώρα, σε σχέση με το Δουβλίνο, και εγώ θα ε, πρότεινα να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές. Εάν θέλουμε να ληφθεί απόφαση, τότε και θέλουμε επίσης τα κράτη-μέλη να μην προβάλλουν αντίσταση, πρέπει ε, είτε να υπάρχει μία πλήρης ανακατανομή, ε, από την άλλη πρέπει επίσης και να υπάρχουν και ανοιχτές πόρτες, να υπάρχει προθυμία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταλαβαίνει ότι ε, τα κράτη-μέλη έχουν, ε, έχουν αναλάβει εθελοντικά την ε, υποδοχή, την φιλοξενία, την ανακατανομή των ε, προσφύγων. Αυτός ο μηχανισμός ανακατανομής δεν πρέπει να είναι όμως προαιρετικός, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως έχει. Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι δεν έχουν δεχτεί όλα τα κράτη-μέλη αυτό, ε, αυτόν τον ε, μηχανισμό. Ακόμα και σε περίοδους ειρήνης που δεν, δεν, τρέχει, δεν συμβαίνουν και πολλά και πάλι το Δουβλίνο δεν έχει αποβεί αποτελεσματικό. Φανταστείτε τώρα που υπάρχουν κράτη που βρίσκονται υπό πίεση, ε, πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Για αυτούς τους λόγους Πιστεύω πως δεν γίνεται να είναι προαιρετικός αυτός ο μηχανισμός, αλλά να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν και εκείνα ε, με τη σειρά τους. Διαφορετικά, ναι, θα υπάρχει ε, δυσπιστία ή θα υπάρχουν αντιδράσεις. Επίσης, ε, θα ήθελα να προτείνω και πάλι ρεαλισμό. Δεν γίνεται όλα τα κρατημέλη να προτείνουν τα ίδια ε, ιδανικά ε, πρότυπα διαβίωσης. Πρέπει να δούμε επίσης και τι γίνεται στο κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, τις ιδιαιτερότητες, το, ε, τους πολίτες, πώς αντιλαμβάνονται την κατάσταση. Υπάρχει η Γερμανία, υπάρχει η Σουηδία, χώρες που είναι οικονομικά ισχυρές. Υπάρχουν όμως και κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Είναι λοιπόν δύσκολο να εφαρμοστεί εξίσου ένας ε, μηχανισμός. Γι' αυτό λοιπόν ε, όταν ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτόν τον μηχανισμό συγκέντρωσης θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται προσοχή διότι δεν πρέπει να υποπέσουμε σε λάθη και να διευκολύνουμε τους διακινητές. Πρέπει να ξέρουν ότι κάθε πρόσφυγας ο οποίος φτάνει εδώ ε, είτε μέσω, μέσω του οργανωμένου εγκλήματος θα... Ε, μάλλον πρέπει να μην δώσουμε κανένα περιθώριο ε, στους διακινητές. Επίσης, πρέπει να γίνει επιτέλους λόγος για όλα τα ατυχήματα που έχουν συμβεί και όλα, όλους τους ανθρώπους και τις ζωές που έχουν ε, χαθεί στα χέρια των διακινητών. Έχουμε τους τελευταίους τρεις ομιλητές. Η ε, κυρία Βαλέρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω τα υποθέντα. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα. Θα ήθελα να θέσω κάτι το οποίο με προβληματίζει. Ακούσαμε αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι πρέπει να εργαστούμε γρήγορα να καταλήξουμε συγκεκριμένη πρόταση. Έχουμε μια νομοθεσία. Αναφερθήκαμε στη διαδικασία για το άσυλο, στην οδηγία περί υποδοχής είναι νομοθεσίες που χρειάστηκαν κάποιο χρόνο για να προταθούν, να αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων, να εγκριθούν και εδώ και στο Συμβούλιο και μετά όλα αυτά θα πρέπει να σωματωθούν, στα εθνικά κοινο... Ε, να σωματωθούν στις εθνικές ενόμες τάξεις. Εμείς στη Σουηδία εργαστήκαμε, επεξεργαστήκαμε την οδηγία ε, του ασύλου για να στοματώσουμε στην ομοθεσία μας για να μπορέσουμε να κινηθούμε επ' αυτής αργότερα. Και προσπαθήσαμε να μην επιδεινώσουμε τις συνθήκες που ήδη επικρατούσαν στη Σουηδία λόγω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η οδηγία, ε, η φιλοσοφία ήταν πάντα να βελτιώνουμε τους κανόνες από τους προηγούμενους. Αντί να μειώνουμε το επίπεδο της νομοθεσίας είναι κάτι που διαπνέει όλη τη συζήτηση πιστεύω, να καταλήξουμε στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, δηλαδή να κάνουμε λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε. Φοβούμε ότι αν επιταχύνουμε τη διαδικασία, αν θεσπίσουμε μια νομοθεσία βιαζόμενη, δεν θα εξετάσουμε σωστά τις συνέπειες. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος επί της νομοθεσίας των διαφόρων κρατών μελών διότι εφαρμοστικός κανονισμός ε, θα υλοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε να έχουμε καλό επίπεδο, να έχουμε ποιοτική νομοθεσία. Πώς θα μπορέσουμε να την συνδέσουμε με το εθνικό δίκαιο ε, μέσω διεργασιών που θα λάβουν χώρα στα εθνικά κοινοβούλια. Εγώ φοβάμαι τη βιασύνη. Είδαμε με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας Εγκρίθηκαν πολύ γρήγορα οδηγίες και κανονισμοί για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Αλλά άμα κινούμεθα γρήγορα δεν εξετάζουμε τις λεπτομέρειες. Χρειαζόμαστε νομοθεσία που να κρατάει για χρόνια στο μέλλον και όχι μόνο να μπορεί να ισχύει για ένα-δύο χρόνια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που τήρησε το χρονοδιάγραμμα. Presidente, Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σχετικά με τον νέο κανονισμό πρέπει και μπορούμε να αποφύγουμε το μεγάλο σφάλμα ότι ορισμένες μόνο χώρες τελικώς καθίστανται υπεύθυνες για, για τον χειρισμό όλων των θεμάτων του προσφυγικού. Αυτά τα spot από την άλλη μεριά πάνε να γίνουν ανοιχτέ φυλακέ. Στα ίδια μας τα σύνορα, στα, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται να προσφέρουμε τη δυνατότητα υποδοχής ανδρών, γυναικών, παιδιών. Και το Δουβλίνο πρέπει να έχει μια δεύτερη επιλογή. Και σε αυτή τη δεύτερη επιλογή, αυτή να περιλαμβάνεται δηλαδή, και εκεί όπου πρέπει να ε, δειχθεί αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών, για την ώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση, δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση μεταξύ των χωρών. Η υπόθεση αυτή θα συνεχιστεί. Βεβαίως το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία με την Τουρκία για την επανεισδοχή προσώπων που θεωρούμε ότι πρέπει να επιστραφούν στην Τουρκία. Όμως και κάτι άλλο. Έλαβε και την πολιτική απόφαση το Συμβούλιο να επιβάλλει με ακραίο τρόπο την συνθήκη του Δουβλίνου. Και γι' αυτό λέω ότι τα hotspot είναι ανοιχτές φυλακές. Μας λένε οι εμπειρογνωμονές ότι αυτό που θα γίνει είναι ότι απλώς θα αλλάξουν οι οδοί που ακολουθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, διότι αυτοί θα συνεχίσουν να έρχονται και θα χαθούν και άλλες ανθρώπινες ζωές. Γιατί δεν κάνουμε όπως έκανε ο Καναδάς. Λαμβάνουμε μια απλή απόφαση ότι κάθε χώρα μέλος θα υποδεχτεί έναν αριθμό προσώπων. Νομίμως, τότε δεν θα χρειαστεί κανένας να διακινδυνεύει, να κινδυνεύει η ζωή του δηλαδή. Οι δε αιτήσει ασύλου μπορούν να λαμβάνονται και ε, να γίνονται αντικείμενο επεξεργασία στις προξενικές αρχές. Διότι αυτές είναι και που γνωρίζουν καλύτερα τις εθνικές νομοθεσίες των χωρών. Και δεν θα δώσουν τις προξενικές τους θεωρήσεις, θεωρήσεις κατά τρόπον αυθαίρετο. Αυτό νομίζω θα ήταν το κλειδί για την ε, κατάσταση Η ασφαλής δίωδος το secure transit δηλαδή στα αγγλικά είναι αυτό που είναι αναγκαίο για να σταματήσουν να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Προ 80 ετών η μητέρα μου ως μικρό κοριτσάκι ήταν πρόσφυγας πολέμου και σχεδόν πνίγηκε ε, και για να φτάσει μέχρι ε, την χώρα μας. Και ε, μάλιστα έπαθε και τη φοηδή ε, πυρετό και δεν θα ξεχάσει ποτέ τις εμπειρίες αυτές. Ευχαριστώ. Κυρία Βίνμπεργκ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σας πληροφορίες. Πρέπει να πω, δεν είναι ότι δεν κατανοώ τα όσα υπόθηκαν. Μιλήσαμε για νόμιμες διόδους αφήξεως. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε η γαλάζια κάρτα. Ποτέ δεν ήταν επιτυχή η γαλάζια κάρτα. Ήταν απλώ διακοσμητική φύσεω, θα έλεγα. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτή τη λύση και πολύ. Τα κράτη-μέλη ε, και ελληνική μεταξύ τους. Αυτά κουβεντιάζουμε. Πρέπει να δούμε πόσα άτομα πρέπει να ανακατανεμηθούν και πόσα θα τα καταφέρουμε. Θα καταφέρουμε 60.000, θα τα καταφέρουμε εγώ νομίζω μόνο ε, κάνα δύο εκατοντάδες τα καταφέραμε. Κάποιες χώρες λένε ότι δεν ενδιαφέρονται. Δεν θα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό που οφείλουν. Πάντα ζητούσαμε να το κάνουν, να ανταποκριθούν στην υποχρέωση αναδιανομής, ανακατανομής και μετεγκατάστασης. Δεν ξέρουμε πόσοι θα πρέπει να ανακατανεμηθούν, αν δεν ξέρουμε πόσα κράτη-μέλη διαθέσιμα να δεχτούν πρόσφυγες. Χρειάζεται μια ισότιμη κατανομή. Μιλήσαμε και για την ένταξη των ανθρώπων αυτών που θα έρθουν στα κράτη-μέλη. Στη Σουηδία έχουμε μεγάλο πρόβλημα ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων. Πρέπει να δούμε αυτό το παράγοντα. Διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο καταβλισμό, χωρίς ένταξη όπως συνέβη σε εμά. Οι πολίτες στα διάφορα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να τοποθετηθούν επ' αυτού του θέματος μέσω δημοψηφίσματος, να πούν τι θέλουν. Τα κράτη-μέλη που δεν συμφωνούν με μια υποχρεωτική ανακατανομή, τι θα κάνουμε αυτά τα κράτη-μέλη, αν μέλος πει όχι. Πώς θα πρέπει να κινηθούμε, τι θα πρέπει να κάνουμε. Η Έλλη έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Συμφωνώ, λέει η Ελισλάιν, με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Θέλουμε μεγαλύτερο θάρρο να έχει η Ενεκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια στεναρή θέση. Και όχι να παρουσιάζει εναλλακτικέ. Οι εναλλακτικέ δεν είναι ίδιε, δεν είναι ουδέτερε. Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Ε, κάνει τη διαφορά ποια θα συμπεριφθεί στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο η δεύτερη επιλογή οδηγεί σε τολμηρή μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου αντί διακοσμητικές αλλαγές. Και μόνο αυτή την επιλογή θέλουμε. Αναφέρεται ότι είναι νεκρό το Δουβλίνο και πρέπει να ξεπεραστεί, ότι δεν λειτουργεί. Και μετά θα ικανοποιηθούμε λέγοντας αυτό με ένα Δουβλίνο συν ε, η προσέγγιση μέχρι τώρα δεν είχε πετύχει. Οι αριθμοί δείχνουν ότι 6 από τα 28 κράτη-μέλη μόνα τους ε, καλύπτουν 80% των αιτήσεων ασύλου. Στο Κοινοβούλιο τρεις φορές ψηφίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία την ανάγκη να ξεπεραστεί η προσέγγιση του Δουβλίνου. Η ολιστική ε, προσέγγιση στη μετανάστευση και στη δυτική έκθεση που ψηφίστηκε οδηγεί σε επιμερισμό των ευθυνών Ζητά να ξεπεραστεί το κριτήριο της πρώτης χώρας άφηξης. Ζητά τα κριτήρια να θεσπίζονται βάσει του μηχανισμού μεταγκατάστασης, βάσει των συνηθισμένων κανόνων. Και κινείται προς την επιλογή 3. Κεντρικό σύστημα επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου, που θα είναι ευρωπαϊκής ευθύνης. Συμφωνώ με τι ανησυχίε συναδέλφων. Χρειάζεται εναρμόνιση του συστήματος όχι εις βάρος όμως των δικαιωμάτων των ανθρωπίνων. Να μην μειώνεται η προστασία. Πάντα αποτύχανε αυτή η προσέγγιση. Ελπίζω να μην ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τους εγωισμούς των κυβερνήσεων κρατών μελών, γιατί κάτι τέτοιο θα υπονόμευε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Ευχαριστώ. Ελείς συνάδελφοι, θα παρατηρήσατε ότι είμαστε απελπιστικά καθυστερημένοι χρονικά και έχουμε άλλο ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη, το θέμα του Eurojust, εδώ είναι ομιλητές που κάποιοι ήρθαν ειδικά για αυτό το θέμα. Εγώ αναλαμβάνω τις ευθύνες για την πολύ κακή εξέλιξη των εργασιών από πλευράς χρονικής. Θα ήθελα να ακούσω όλες τις παρεμβάσεις των εισηγητών, παράδειγμα. χάρη. Ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει τις παρεμβάσεις. Δεν ήθελα να ξεπετάξουμε το θέμα. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ικανοποιητικό. Θεωρώ ότι άκουσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτά που έθηκαν ήταν πολύ ευφυή, ε, ε, εκφράστηκαν με πάθος αρκετοί από τους ομιλητές και ελπίζω να τα έλαβε υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει νόημα να απαντήσετε σε όλα αυτά τώρα, δεν έχουμε χρόνο. Και κύριε Σκέμπρη, ελπίζω να σημειώσατε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Αποφάσισαν να ακουστούν όλοι. Κάθε συνεισφορά ήταν σημαντικότατη σήμερα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Σημείωσε δεόντως τα υποθέντα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις μελλοντικέ συζητήσεις θα εστιαστούμε επί λεπτομεριών της ανακοινώσεως και άλλων συναφών λεπτομεριών για τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Ευχαριστώ για την υπομονή σας, συνάδελφοι. Πάμε τώρα στο σημείο 9 παρουσίαση από την Eurojust. Η πρόσωπος της Eurojust δεν έχει την καλοσύνη η Μισελ Κόνιξ να έρθει εδώ. Πάμε αμέσως σε αυτό το σημείο, συνάδελφοι, για να προχωρήσουμε. Θα ξεκινήσω την εισαγωγή στο θέμα ενώ καταφτάνει η Μισελ. Um, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε λοιπόν την παρουσίαση σε πλευρά τη Μισελ Κόνιξ, τη Προέδρου του Eurojust, που θα παρουσιάσει την τρίτη έκθεση του Eurojust. Θέμα «Οι ούτως αποκαλούμενοι ξέρει, ε, ξένοι συγγνώμη, μαχητές ξένοι τρομοκράτες μαχητές. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων μετά με τα μέλη. Δεν θα κάνω άλλη εισαγωγή λόγω λύψης χρόνου και ζητώ συγγνώμη για τις καθυστερήσεις. Λοιπόν, ακούμε την παρουσίασή σας, Μισελ. Ξεκινήστε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Διακεκριμένα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, τιμή για μένα να παρουσιάσω το έργο του Eurojust στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και εδώ θα αντικατοπτρίζεται και η έκθεση της συνεδριάσεως που ήταν αποτέλεσμα της συνεδριάσεως που έγινε τον Ιούνιο του 2015 εδώ και 10 μήνες περίπου εδώ μεταξύ πολλά συνέβησαν πρώτο σχόλιο κάποια προκατατικά σχόλια έχω αν επιτρέπετε λοιπόν τα θύματα θέλω να αναφέρω. Γι' αυτό εργαζόμαστε τόσο σκληρά. Αδίσταχτα αποτείουμε φόρο τιμή στα θύματα τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και αλλού, σε όλο τον κόσμο, λόγω των θυμάτων, λόγω της προσπαθίας να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσω διώξεως των εκείνων των ενόχων για αυτά τα εγκλήματα. Λόγω αυτής της προσπαθίας αυτής και λόγω των θυμάτων έχουμε κίνητρο να εργαζόμαστε άοκνα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτή η έκθεση είναι συνοπτική έκθεση. Είναι η εκδοχή συνοπτική μιας πιο λεπτομερούς εκθέσεις που βάλαμε στους Υπουργούς Εσωτερικών πέρσι το Δεκέμβριο αυτή η έκθεση που παρουσιάστηκε πέρσι είναι ε, ε, ε, απόρριτη θα έλεγα και εδώ είναι συνοπτική έκθεση. Καρπός αυτή η έκθεση είναι της ανταλλαγής απόψεων ε, εισαγγελέων ειδικευμένων στην καταπολέμηση τρομοκρατίας που διενεργούν έρευνες και διώξεις. Θέλαμε λοιπόν να μάθουμε από τα μαθήματα. Θέλαμε να γίνει ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Τώρα, εάν αποκαλυφθούν τα πλήρη περιεχο... αν αποκαλυφθεί το πλήρες περιεχόμενο των εκθέσεων, ε, θα είναι επικίνδυνο για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, είναι εμπιστευτικό το έγγραφο, μπορώ να αναφερθώ σε γενικές παρατηρήσεις, σε μαθήματα κλπ. και βέλτιστες πρακτικές, αλλά δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες διότι διεξάγονται διώξεις και έρευνες και αν θα ήταν αντιεπαγγελματικό αν αναφερόμουν σε λεπτομέρειες και θα καταστραφεί η εμπιστοσύνη που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τους εισαγγελείς τους υπεύθυνους με καταπολέμηση των τρομοκρατών. Καθοδηγούμεθα θα τα γεγονότα, από τη ζήτηση και θέλουμε όμως στόχος μας να είναι τα αποτελέσματα της εργασίας. Είμαστε οι πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2012 που εντοπίσαμε το πρόβλημα των ξένων μαχητών, των τρομοκρατών αυτών. Και αυτό χάρη στην εμπιστοσύνη που δημιουργήθηκε μετά από τις συζητήσεις δικτύωσης με τους εθνικούς εισαγγελείς, τους υπευθύνου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. NCTs εν συντομία θα τους αποκαλούμε. Συναντηθήκαμε αυτούς το 2012 και τα τελευταία 10 χρόνια τους συναντούμε βάσει τη αποφάσεω του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005. Έτσι υποχρεώνται τα κράτη-μέλη να καθορίσουν εθνικού υπευθύνου για την τη τρομοκρατία και πρέπει να μα ενημερώνουν για αυτά που συμβαίνουν στα κράτη-μέλη σε κάθε φάση ποινικών ε, διώξεων. Και αυτό συστηματικά οδηγεί σε τακτικές συναντήσεις με αυτούς τους ανθρώπους από το 2005 μέχρι σήμερα. Το 2012 ένας από τους NCTs μας ζήτησε να διαπιστώσουμε αν οι ξένοι μαχητέ ήταν εθνικό πρόβλημα συγκεκριμένο. Και χάρη σε ένα ερωτηματολόγιο που απεστάλλει μετά τη συνεδρίαση του Ιουνίου του 2012, Σεπτέμβρη του 2012, ήδη ανακαλύψαμε το έτος αυτό ότι δεν ήταν μόνο μια χώρα, αλλά και άλλες έξι χώρες που αντιμετώπιζαν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή οι υπηκόρους πηγαίνουν στη Συρία, στο Ιράκ και επέστρεφαν, και καμιά φορά επέστρεφαν με τρομοκρατικές προθέσεις και κάποιοι από αυτούς ε, στατολογούσαν όλους, αναμεγνιόταν στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών επιθέσεων και είχαν πρόθεση κάποιοι από αυτούς να επιτεθούν κατά αθών εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αλλού. Και γι' αυτό το 2013 ξεκινήσαμε την συζήτηση για αυτούς τους ξένους μαχητές της συναντήσεις του δικτύου. Περιγράψαμε πέρσι ποια ήταν τα αποτελέσματα της συνεδρία του 2014. Το κάναμε αυτό το 2013, το 2014 και το 2015 σας ενημερώναμε για τα αποτελέσματα. Πριν από τις επιθέσεις που έγιναν το μεταξύ, εξετάζαμε τι πρέπει να κάνουμε να είμαστε αποτελεσματικότεροι στην καταπολέμηση τρομοκρατίας ποιος θα ασχοληθεί με συγκεκριμένο τμήμα της πραγματικότητας για να είμαστε αποτελεσματικοί. Γιατί χρειάζεται κάτι, πότε χρειάζεται κάτι, πώς θα κινηθούμε. Αυτό θα είναι και το πνεύμα της παρουσιάσεως σήμερα. Αν πιστεύετε ότι το Eurojust δίνει στατιστικά στοιχεία, όχι είμαστε δικαστικός φορέας που επιχειρησιακά, τακτικά και στρατηγικά κινείται συναθρίζοντας τους υπευθύνους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 100.000 επιστρέφοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσουμε από αυτούς που πηγαίνουν να πολεμάνε και επιστρέφουν. Τι χρειαζόμαστε δικαστικά, νομικά, στρατηγικά. Ε, είναι περίπλοκο το πρόβλημα. Ένα περίπλοκο πρόβλημα δεν επιλύεται απλά. Είναι δυναμικά μεταβλητό πρόβλημα. Απαιτεί δυναμική προσέγγιση και όχι στατική. Και τι ζητούσαμε πάντα τα τελευταία χρόνια. Κοινή σφαιρική κάλυψη και προσέγγιση. Η δικαστική πτυχή αποτελεί τμήμα της ολιστικής κοινή προσέγγισης. Ένα παράδειγμα. Αν είναι χρήσιμο να τους καταπολεμήσουμε τους ξένους μαχητές φυλακίζοντάς τους, καταδικάζοντάς τους. Αν τους στείλει στη φυλακή, οι φυλακές είναι θύλακες, ε, εποάζονται εκεί τρομοκράτες. Ε, είπαμε ότι καταδίκες για το σκληρό πυρήνα για τους βετεράνους έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Και το είδαμε μέσα, είδαμε την απόδειξη. Όταν μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες ε, είδαμε ότι είπε ένας από τους την άχτηκα, είπε στη διαθήκη του, διότι δεν θέλω να πάω φυλακή. Υπάρχει αποτρεπτικός χαρακτήρας αυτά τα μέτρα της φυλάκησης. Θέλουμε κοινή προσέγγιση, πλήρη προσέγγιση. Άρα πρέπει να εξετάσουμε διάφορα επίπεδα κινδύνου που αντιπροσωπεύουν οι διάφοροι ε, ξένοι μαχητές, ε, διάφορους λόγους για τους οποίους κινούνται, αυτοί που επιστρέφουν αφού πάνε στη Συρία και στο Ιράκ και αναμειγνύονται στις συγκρούσεις στον πόλεμο, επιστρέφουν με τραύματα άλλοι χωρίς τρομοκρατικές προθέσεις. Άρα ε, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι διαφορε... με διαφορετικό ιστορικό, διαφορετικός λόγους, διαφορετικές προθέσεις. Δημιουργούνται επικοινόμορφα, άρα είναι περίπλοκο πρόβλημα που δεν δίνεται απλά. Έχουμε και δικαστική διάσταση, λοιπόν στο όλο θέμα της καταπολεμήσεως των ξένων μαχητών και είναι σημαντικότατη. Τι ζητούσαμε στις τελευταίες εκθέσεις. Κοινό νομικό πλαίσιο θέλαμε και πρέπει να πω ότι λόγω του ψηφίσματος του ΟΗΕ της 21-17 του Σεπτεμβρίου του 2014 λόγω των πρωτοβουλίων του Μαΐου 2015 σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης μέσω του δεύτερου συμπροματικού πρωτοκόλου της Συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη τρομοκρατίας ε, πάρα πολύ σημαντική επίσης που είναι και η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη DG Home που δρομολόγησε τις συζητήσεις περί οδηγίας για κοινό νομικό πλαίσιο. Για όλους αυτούς τους λόγους λέω ότι κινούμεθα προς σωστή κατεύθυνση. Από το 2002 έχουμε απόφαση πλαίσιο που δίνει κοινό ορισμό της τρομοκρατίας. 2008 δείχνησαν τις λεπτομέρειες της αποφάσεως συμπεριλαμβάνοντας αυτήν την στατολόγηση, την εκπαίδευση, την πρόκληση παρακίνηση τη δημόσια. Μετά προσπαθήσαμε ε, να δούμε τι γίνεται με τα ταξίδια, χρηματοδότηση των ταξιδίων. Εάν κανείς ταξιδεύει με τρομοκρατική πρόθεση, τι κάνουμε. Και θέλαμε να εμποδίσουμε τον κόσμο να ταξιδεύει με τρομοκρατική πρόθεση. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την κοινή πτυχή να καταπολεμήσουμε. Είναι καλό ότι τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ούτως ώστε κάτωθεν να κινηθούν θεσπίζοντας την νομοθεσία για να δουν αυτά που τονίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΙΕ τα στοιχεία για την καταπολέμηση της δημοκρατίας. Χρειάζεται κοινή γραμμή από τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η ουσία. Ο λόγος ύπαρξης της οδηγίας. Ζητήσαμε κοινή προσέγγιση. Διότι τι είδαμε, ότι κάποια κράτη-μέλη είχαν υψηλό νομοθεσία. νομοθεσίας. Κάποια κράτη-μέλη δεν είχαν τη σωστή νομοθεσία. Στην τελευταία συνεδρίαση των υπευθύνων για την καταπρόσωση της ότι πολλοί από τους αγγελείς εποφελούνται από πρόσφατες αλλαγές στι νομοθεσία της χώρας τους. Καλωσορίζουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG Home κάλεσε τη Eurojust να συμβάλλει στη συζήτηση να τοποθετηθεί πώς την πράξη θα ωφελούσε η κοινή νομοθεσία. Είχαμε κάποια κενά που διαπιστούσαμε. Κενά διοκτικά. Όταν κάποιος είναι απλώς μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης δεν είναι αρκεί. Η συνεισφορά σου στις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας καθορίζει αν η συμπεριφορά σου χαρακτηρίζεται τρομοκρατική, τι αυτή. Και μετά, βλέποντας την ομολογία, είδαμε ότι κάποιες νέες γυναίκες και παιδιά που ταξίδευαν προς Συρία και Ιράκ και επέστρεφαν εδιώκοντο για τρομοκρατική δραστηριότητα διότι ε, έδωσαν, βοήθησαν με τη μεταφορά διότι μαγείρευαν για τους ξένους μαχητές και βλέπουμε ότι η ίδια συμπεριφορά δεν τιμωρείται σε άλλες χώρες αν τιμωρείται σε άλλες. Σε κάποιες χώρες αντιμετωπίζονται προβλήματα όσον αφορά την παθητική κατάρτιση. Εμείς τιμωρούμε μόνο την ενεργό κατάρτιση. Είδαμε διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά ποινικά στοιχεία ανάλογα με το πώς, αν καλύπτεται ή όχι από την νομοθεσία σου η ριζοσπαστικοποίηση. Είδαμε με την ομολογία ότι κάποια δικαστήρια έστειλαν σαφή μηνύματα Υπήρχε λεπτή διαχωριστική γραμμή από την υπεράσπιση λέγοντας αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Πηγαίνοντας στις περιοχές συγκρούσεων σχετίζεται με τη σύμβαση της Γενέβης με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Είχαμε πολλές καταδίκες από το 2008 και μετά παρακολουθώντας το τι γίνεται αναλύοντας τις καταδίκες πολλές Πολλά δικαστήρια είπαν ότι μια συγκεκριμένη πράξη θεωρείται τρομοκρατική και κάποια συγκεκριμένα κράτη-μέλη προσάρμοσαν δεόντως την ομολογία τους ε, σύμφωνα με την απόφαση πλαίσιο του 2008. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζεις εκείνους που επιστρέφουν, πώς τους ποινικοποιεί. Είδαμε ότι κάποιες χώρες εξέτασαν τον κίνδυνο, δείκτες κινδύνου, έκανα αξιολόγηση κινδύνου, αποτίμηση κινδύνου και θεώρησαν ότι είναι πολύ επικίνδυνοι αυτοί που επιστρέφουν. Ανάλογα, ε, επιστρέφονται σε υψηλού επικινδύνου, μέσου χαμηλού κινδύνου. Ε, και έγινε ανταλλαγή πρακτικών για να δουν κατά πόσο μια χώρα ήθελα να μιμηθεί την άλλη ε, όσον αφορά αυτή, αυτό το διαχωρισμό. Χρειάζεται όμως σωστό νομικό πλαίσιο, δικαστικό πλαίσιο, να καθορίσουμε τι θεωρείται επικίνδυνο. Ε, ποιος ο λόγος που κατονομάζεις κάτι με έναν τρόπο ή όχι. ποιο είναι ο κίνδυνος από τη μετακίνηση. Από την εμπειρία λοιπόν με τους SETs είδα ότι πρέπει να προσέξουμε τους σκληρού βετεράνου, αυτοί που πήγαιναν Με, ε, και αυτούς που έχουν ιστορικό ε, μητρό έχουν κάνει αδικήματα απλά, αν θέλετε, εγκλήματα, σοβαρά εγκλήματα και τρομοκρατικά εγκλήματα. Αρέθεσα κάποια παραδείγματα. Ο Αντελαχήμ ερήμην είχε καταδικαστεί τον Ιούλιο, 20 Ιουλίου, που αδικαστεί των Βρυξελών. Άλλος καμικάζει στις επιθέσεις των Βρυξελών, καταδικάστηκε από το ίδιο δικαστήριο και άλλους Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα λαμβάνουμε υπόψη δικαστικός πώς και θέλουμε και από ρίζοσπαστικοποίηση να επιδιώκεται. Προδικαστικά κατά τη διάρκεια της ε, δίκης και μετά τη δίκη και κατά περίπτωση εξακριβώνουμε σε ποιο στάδιο, σε ποιο βαθμό μπορεί να αλλάξει κάπως ε, η δίωξη και να ζητήσουμε εναλλακτικέ κυρώσει. Το Συμβούλιο μετά τη διάσκεψη της οποίας ηγήθηκε η Τζούροφα στις 9 Οκτωβρίου του 2015 αποφάσισε να αναθέσει στο Eurojust την παρακολούθηση των διαφόρων προγραμμάτων από όριζες πρακτικοποίησης πριν τις δίκες και μετά τις δίκες. Αλλά και αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να σκεφτούμε τα προγράμματα απορριζοσπαστικοποίησης βάση κοινοτήτων και μετά να κυνηγήσουμε τα αίτια, τη ρίζα του κακού. Τώρα, να επιστρέψω και σε κάτι άλλο. Την ανάγκη για τα στοιχεία, ψηφιακά στοιχεία, που τα χρησιμοποιούν εκτεταμένα οι τρομοκράτες μέσω διαδικτύου και κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Και έχουμε προβλήματα για να μαζέψουμε στοιχεία, αντιμετωπίζουμε προβλήματα λόγω Τη οδηγία για την προστασία, για τη συντήρηση των στοιχείων, διατήρηση των στοιχείων και αυτό διότι υπάρχουν διάφορα συστήματα για την προστασία δεδομένων στα διάφορα κράτη-μέλη. Επίση, βλέπουμε ότι η δικαστική συνεργασία με τρίτες χώρες είναι σημαντικότατη. Εργαζόμεθα πολύ πάνω σε αυτό το τομέα για τη δικαστική συνεργασία και πολλά ακόμα θα κάνουμε. Περιμένουμε ερωτήσεις. Αν προλάβουμε, αν προλάβουμε. Η κυρία Χολμάιρ έχει το λόγο. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Η Επιτροπή μας έχει με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για τις γενικές εκατευθύνσεις που έχετε λάβει. Ε, καταλαβαίνω και όλα σε αυτό που μας είπατε ότι δεν μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις ε, τρέχουσες έρευνες. Ε, έχω απόλυτη κατανόηση σε αυτό. Ε, θα είχα κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα συμπεράσματα. Καταρχάς, βλέπω ότι υπάρχει ισχυρή ε, σχέση της τρομοκρατίας με το πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τους ξένους μαχητές ε, στον ε, τομέα τον ε, ποινικό. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ποινικό δίκαιο. Πιστεύω πως αυτό είναι ένα αρκετό, αρκετά σημαντικό ερώτημα. αρκετα σημαντικο από την άλλη, στην έκθεσή σας αναφέρετε ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να έχουμε πληροφορίες για τα ταξίδια με τρομοκρατικές προθέσεις. Ε, έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση και ε, με, τα ταξίδια, να μην απαγορευτούν τα ταξίδια γενικότερα, αλλά τα ταξίδια με προθέσεις τρομοκρατικές και εάν υπάρχουν ε, διασυνδέσεις με κάποιο τρομοκρατικό δίκτυο ή με κάποια τρομοκρατική ενέργεια. Είναι, πιστεύω, όντω πάρα πολύ σημαντικό. Έπειτα, σε σχέση με την εκπαίδευση, εδώ υπάρχει μεγάλη επισφάλεια. Ακούσαμε και χθε από έναν Ιταλό εισαγγελέα ότι όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις ε, έρευνες ε, για τη ρίζοσπαστικοποίηση, μας είπε ότι παρατηρούνται υψηλά ποσοστά ριζοσπαστικοποιημένων Ισλαμιστών, ότι υπήρχε μέχρι και ένα πεντάχρονο κοριτσάκι σε ένα ε, βίντεο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης και πολύ πιο σημαντικό μάλιστα όταν έχει να κάνει με παιδιά. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά και να αποτρέψουμε την κακομεταχείρισή τους, κακοποίησή τους από τους ίδιους τους, τους γονείς. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τα όσα μας είπατε για την άπορη ζωσπαστικοποίηση. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τις βέλτιστες δυνατότητες και τα ε, σωστά μοντέλα άπορη ζωσπαστικοποίησης. Ιδιαίτερα τα μέτρα μπορούν να ληφθούν μέσα στις φυλακές για εκείνους που έχουν ήδη καταδικαστεί και δεν έχουν καμία απολύτως ε, προοπτική και σαπίζουν πίσω από τα σίδερα υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, από ριζοσπαστικοποίησης ακόμα και για ε, αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να αρχίσει η διαδικασία από ριζοσπαστικοποίησης ήδη μέσα από τις φυλακές. Καθώς επίσης και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξερευνήσουμε το δυναμικό της Eurojust, να συνδυαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μας δώσουν αρκετές ε, πληροφορίες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το νομοθετικό μας έργο. Από τη μία πιστεύω πως ε, σίγουρα είναι χρήσιμη μια οδηγία που να αναφέρεται στο ποινικό δίκαιο και να υπάρχει εναρμόνιση νομοθεσίας. Από την άλλη όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την απορριζοσπαστικοποίηση, τα οποία θα πρέπει φυσικά να, να ψηφίσουν τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέρκοπ έχει το λόγο. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Καταρχάς, η φιλοδοξία που υπάρχει για εναρμόνιση ποινών και ε, περιγραφής αδικημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω πως δεν μπορούμε να κάνουμε τη φιλοδοξία πράξη. Ωστόσο, Φαίνεται ότι κάποιες από τις προτάσεις σας για τεχνικά πρότυπα, τα οποία αφορούν ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, έχουν ε, πολύ περισσότερες πιθανότητες να πραγματοποιηθούν. Είναι πιο εφικτά. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει αυξημένη συνεργασία. Υπάρχει το έκρηση, υπάρχει το σύστημα PNR ε, και όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Γι' αυτό πιστεύω πως θα έπρεπε ίσως εκεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Ορισμένες φορές δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά ε, συμβάντα, ιδιαίτερα στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών, ακριβώς επειδή ε, διαφέρουν τόσο πολύ τα τεχνικά πρότυπα από χώρα σε χώρα. Και Δεδομένου τούτου θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας για τη συνεργασία ανάμεσα στις ε, υπηρεσίες. Αναφέρατε τη Frontex, τη Eurojust και τη Europol και είναι σίγουρα ζωτική σημασία. Υπάρχει όμως ε, μία πληθώρα άλλων υπηρεσιών που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν μέσω της συνεργασίας. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, κοινέ ομάδες ερευνών. Είδαμε στο παρελθόν ότι Υπήρχαν πολλές ευκαιρίε για κοινέ επιχειρήσεις, ωστόσο τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Δεν έγινε τίποτα ή μάλλον δεν έγιναν και πολλά. Έχουμε δει επίσης ε, αρκετές επιτυχίες στις περιπτώσεις όπου έχει υπάρξει συνεργασία. Και ίσως θα έπρεπε να κοιτάξουμε το ενδεχόμενο μιας αναθεώρησης, διότι ίσως βελτιωθεί η μαλλον δεν εγιναν και πολλα εχουμε δει επισης αρκετες επιτυχιες στι περιπτωσεις οπου εχει υπαρξει συνεργασια και ισως θα επρεπε να κοιταξουμε το ενδεχομενο μιας αναθεωρησης διοτι ισως βελτιωθει η κατασταση να δούμε εάν υπάρχουν λήψεις, προβλήματα ή εμπόδια τα οποία ε, εμποδίζουν στο να χρησιμοποιήσουμε ευρύτερα τα JETs. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρισπέκ. Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου επιθυμώ να ευχαριστήσω την ε, κυρία Διευθύντρια για την θαυμάσια πραγματικά ανάπτυξη του θέματος για ένα θέμα που όπως εξήγησε είναι επίκαιρο εδώ και πολλά χρόνια και πριν ακόμη από τις φρικαλές και αποκλειστικές επιθέσεις που έζησε η Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Άρα ένα θέμα τόσο σοβαρό και ένα προβληματισμό με τόσες διακλαδώσεις και τόσο τρομερό που εσείς περιγράψατε με ρεαλισμό αλλά και ακρίβεια. Ε, τονίσατε βεβαίως και την ανάγκη εμπιστευτικότητας και υπενθυμίσατε, αλλά τα γνωρίζω και εγώ προσωπικά αυτά, την κατάσταση των θυμάτων, των θυμάτων κατά πρώτης των λόγων και των οικογενειών τους. Μέσα από την ε, παρουσίασή σας αντιλαμβάνεται κανείς περισσότερα και από τις ε, λεπτομέρειες ότι τα ε, συστήματα αυτά δημιουργούν δίκτυα, δηλαδή τα τρομοκρατικά δίκτυα και ότι επομένως τους επιτρέπει να δρουν με ταχύτητα ε, όπως είπα, μέσα σε δίκτυα, δικτυώνονται με όλες τις ε, πρόσφορες σύγχρονες τεχνολογίες και δείχνει επίσης και πόσο είναι αναγκαίο να συνεργαστούν πολύ στενά οι χώρες μέλη με ανταλλαγή πληροφοριών που ελπίζω κάποτε να μπορεί να γίνεται σε πραγματικό χρόνο και με πραγματικά αποτελεσματικό τρόπο. Ιδίως όμως πόσο σημαντικό είναι να θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο που να μας επιτρέπει να κινούμεθα ταχαίως και τελικώς να έχουμε το πάνω χέρι σε αυτόν τον πόλεμο ή σε αυτή τη μάχη αν θέλετε. Δύο ερωτήσεις σύντομες μετά από τα όσα εξηγήσατε. Μιλήσατε για έξι χώρες που αφορώνται από τους αλλοδαπούς μαχητές. Ποιες είναι αυτές. Εγώ είχα την αίσθηση ως Ευρωπαία ότι θυγόμαστε όλες οι χώρες, ίσως σε διαφορετικούς βαθμούς. Δεύτερη ερώτηση, πάλι της ευρωπαϊκής επικαιρότητας, έχουμε τη νέα οδηγία για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Ποια είναι η άποψή σας για την ε, πρόταση αυτή, ποιες είναι οι παρατηρήσεις και ενδεχομένως οι προσθήκες που θα θέλατε να δείτε να γίνονται αναπτύξτε μας την άποψή σας σε σχέση με αυτό το σημαντικό κείμενο, έτσι ώστε προϊόντος του χρόνου να καταλήξουμε σε ένα κείμενο, διότι αφοσιώνουμε πολλή ενέργεια για την αναθεώρηση των κειμένων που επεξεργαζόμαστε και κάποιες φορές μετά από ορισμένου μήνες χρειάζονται επανεξέταση. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η οδηγία και είναι σημαντικό επίσης να την ε, ε, φτιάξουμε έτσι ώστε να είναι αποδοτική. Ευχαριστώ κύριος Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση κυρία Διευθύντρια. Ερωτήσεις σχετικά με τα συμπεράσματα που εξάγεται από τις εργασίες σας. Αφενός, από τις υποθέσεις που επεξεργάζεστε έχει την ικανότητα, έχει τη δυνατότητα αν θέλετε να διαπιστώσετε ότι η τρομοκρατία αρχίζει και διασυνδέεται περισσότερο και με το κοινό ποινικό έγκλημα και όχι μόνο σε ό,τι αφορά την παράνομη διακίνηση προσώπων αλλά και για παράδειγμα στο βρώμικο χρήμα. Βεβαίω, εστιάζουμε τώρα περισσότερο στην τρομοκρατία. Σας προκαλεί αυτό την αίσθηση ότι χρειαζόμαστε κάποια εξισορρόπηση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον ορισμό της τρομοκρατίας και αν ανοίγονται εκεί κάποιες δυνατότητες στενότερη συνεργασίας. Τρίτος τομέας, τουλάχιστον έχει κανείς όλο και περισσότερο την αίσθηση ότι στις χώρες μας αυτό θεμελιώνεται περισσότερο. Δηλαδή εξηγώ, έχετε την εντύπωση ότι υπάρχουν ξεκάθαρες δομές μέσα στο εσωτερικό των χωρών μελών. Τα γνωρίζουμε λίγο από την χώρα μου, την Γερμανία, όπου κυριαρχούν σε ορισμένες περιοχές αραβικές συμμορίες, ας το πω εντός εισαγωγικών, προσπαθώντας να μεταφράσω ε, στα ελληνικά τα, την ε, ε λέξη clans. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την παρουσίασή σας που μου φάνηκε σημαντική και επίκαιρη και δείχνει πόσο χρειαζόμαστε ε, συγκεκριμένη και επίκαιρη γνώση. Πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι ο ISIS. Πρόκειται για μια κίνηση, για μια οργάνωση η οποία διεξάγει πόλεμο κατά πολλών από τις χώρες μας. Συμμετέχει σε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις. Όταν ε, κάποιος ξεκινά από ευρωπαϊκή χώρα για να στρατευτεί στον ISIS, αυτό αποτελεί προδοσία κατά της χώρας του. Για να αντιμετωπιστεί αυτό όμως χρειάζονται και οι απαραίτητες νομικές βάσεις. Όταν κάποιος στρατεύεται σε τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις, είτε ως μαχητής είτε και παρέχοντας υποστήριξη χρηματική ή ε, υλική, αυτό όπως είπα χρειάζεται αντιμετώπιση. Δεν είναι απαραίτητο να είναι άκαμπτο το νομικό πλαίσιο, μπορούν να προβλέπονται ενδεχομένως και εναλλακτικέ κυρώσεις όπως είπατε, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρξει η σωστή κατεύθυνση. Αυτό αντιμετωπίζουμε de facto. Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Και οφείλουμε να δούμε τους ανθρώπους αυτούς ως εχθρούς των χωρών μας. Εφόσον κάποιο πρόσωπο δραστηριοποιείται εχθρικά απέναντι σε μια χώρα, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να απελάβνεται από τη χώρα αυτή. Για παράδειγμα, εφόσον κάποιο πρόσωπο διαθέτει διπλή υπηκότητα και στρατεύεται σε μια ε, ε, τρομοκρατική οργάνωση, πρέπει να μπορεί να το αφαιρεθεί η μία ηθαγένεια. Αυτό είναι μια πρακτική λύση. Δύσκολη μεν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εξεταστεί. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ εξωτερήκευση συναισθημάτων κλπ. Με ενδιαφέρει το κοινωνικό γίγνεσθε. Απέναντί μας έχουμε συχνά και ασαφή μηνύματα. Μιλούμε για ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί όμως στην τρομοκρατία. Γι' αυτό και οφείλουμε να εξετάσουμε. Ριζοσπαστικοποίηση σημαίνει, για παράδειγμα, ενεργό υποστήριξη της τρομοκρατίας. Χρειάζεται να εξεταστούν αυτά τα πράγματα και κοινωνιολογικά. Και μάλιστα να προλαμβάνεται η ριζοσπαστικοποίηση. Χρειάζεται να παρακολουθούμε τις ε, απόψεις που εκφράζονται. Αυτό είναι και μια από τις πτυχές του ISIS. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να αποκλειστούν από τις κοινωνικές δομές εφόσον διαβιούν στις κοινωνίες μας. Υπάρχουν και λόγοι να ενταχθούν στις κοινότητες και στις κοινωνίες μας. Αλλά η απομόνωση αυτών οι οποίοι δεν επιθυμούν να διαβιώσουν ειρηνικά μέσα στις κοινωνίες αυτές είναι επίσης αναγκαία. Ευχαριστώ τζεντίνη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτη. Μιλήσατε για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και για εναλλακτικού τρόπους. Μπορείτε να επεκταθείτε λίγο. Δεύτερο, μιλήσατε για την ποινικοποίηση των μετακινήσεων, των ταξιδιών. Διερωτώ είναι ο σωστός τρόπος να κινηθούμε, δηλαδή ποινικοποίηση της πρόθεσης, της εκπαίδευσης, αλλά μήπως προκαλούμε σημαντικές παρενέργειες αν αρχίσουμε τώρα να ποινικοποιούμε τα ταξίδια. Εγώ γνωρίζω σύρους που τους επέτρεψαν τελικά να επιστρέψουν στο κουρδικό τμήμα της Συρίας μετά από μια δύσκολη ζωή στην Ευρώπη και ο τρόπος με τον οποίο μετακινήθηκαν είναι ο ίδιος, οι ίδιες οδοί, οι ίδιοι τρόποι με τους τρομοκράτες. Αν αρχίσουμε να ποινικοποιούμε τα ταξίδια αυτά, πού θα βγούμε. Έχετε σκεφτεί τις παρενέργειες. πει μαχητές να αχθούν ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστήριων. Μάλιστα, ναι, ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Όμως, σε τι θα βασιστούμε για να αποδείξουμε ότι κάποιος αγωνίστηκε στις τάξεις του ΝταΕΣ. Θα σας αρκίσουν κάποιες πηγές από υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών ή θα αναζητήσετε και άλλες πηγές. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ξαναδίνω το μικρόφωνο στην κυρία Κόνιξ, αλλά πρώτα να ρωτήσω για την ριζοσπαστικοποίηση, όπως είπαν και οι κυρίες Χόλμαρ και Σαρτζεντίνη. Ερώτηση λοιπόν, πολύ ειλικρινός, ο Ευρωτζάστ αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Πολλές άλλες, πολύ, ε, συγγνώμη, πολύ λίγες άλλες οργανώσεις έχουν ε, τολμήσει να προχωρήσουν στην ε, ε υπόθεση αυτή. Υπάρχει πραγματική κρίση εδώ. Μιλούμε δηλαδή για αριθμούς ατόμων και πυρήνες που προχωρούν σε ακραία τζιχαντιστική ριζοσπαστικοποίηση. Υπάρχουν όμως νομοταγείς Ισλαμικές κοινότητες και αυτό τη στήριξε βαριά. Πρόκειται για σημαντική κρίση. Από την σκοπιά του Eurojust Βλέπετε κάποια ας πούμε διασύνδεση μεταξύ των πολύ, πώς να πω, ε, περιορισμένων απαντήσεων που δίνουν οι ε, Θα τα ξέρει αυτά ο κ. Κύρκοπ, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αντιδρά με καλές προθέσεις μεν, αλλά η εφαρμογή των μέτρων είναι πραγματικά πάρα πολύ περιορισμένη. Ε, ειδικά δηλαδή ε, για την εκπαίδευση των δασκάλων και το καθεξής. Η Eurojust γνωρίζει πόσο άσχημα προσαρμοσμένες είναι οι απαντήσεις ε, στα προβλήματα αυτά και σε ό,τι αφορά αυτούς που επιστρέφουν. Κάθε χώρα μέλος έχει κάνει διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει μια πραγματική συνοχή ανάμεσα στις αγγελικές διώξεις και στις άλλες ε, απαντήσεις, παρόλο που γνωρίζω ότι κάνετε μεγάλη προσπάθεια για να αποκαταστήσετε μια συνοχή. Υπάρχει όμως κάποια συνοχή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αυτοί που επιστρέφουν. Θα ξεκινήσω από την ερώτησή σας κύριε Πρόεδρε. Πράγματι υπάρχει απειλή για την ασφάλεια και σοβαρή ανευπροηγουμένου απειλή για την ασφάλεια. Θα πρέπει να την πάρουμε στα σοβαρά. Ξεκινήσαμε λοιπόν τις εργασίες μας ε, επί του φαινομένου το 2012. Ε, θεωρήσαμε ότι είναι σαν πετρελοκυλίδα. Έξι χώρες το 2012, ερχόμενοι στην ερώτηση Γείας Γκρισμπέκ το 2012, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ε, αυτές οι χώρες έπρεπε να αντιμετωπίσουν τους ξένους μαχητές, να μην ξεχνούμε την ευρηματική δίκη στην Ανβέρσα τον Φεβρουάριο του 2015 κατά 46 μελών Σαρία for Belgium της, ε, που στατολογούσαν. Η παρουσία του Σαρία for Belgium είχε τεράστια επιρροή στις εργασίες μας όσον αφορά τα δίκτυα στατολόγησης για αλλοδαπούς μαχητές στο Βέλγιο και μετά η συνέχισε να μεγαλώνει. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση εκαλύφθη όχι μόνο 6-7 αρχικές χώρες, αλλά είδαμε ότι όλοι αποτελούν ένα κομμάτι του χάρτη και βλέπουμε βλέπε διαφορές μεταξύ χωρών, βλέπουμε ε, διαφορά όσον αφορά την πυκνότητα του πληθυσμού, του μουσουλμανικού πληθυσμού που είναι παρόν, αλλά δεν μπορούμε να στιγματίζουμε ε, τους μουσουλμάνους που είναι και αυτοί θύματα και θα πρέπει να προστατεύονται. Και γι' αυτό τα κάνουμε όλα αυτά. Για να προστατεύσουμε τα θύματα. Να αποδοθεί δικαιοσύνη. Υπάρχει μεγάλη κρίση πραγματική. και η δουλειά του Eurojust που δεν θα δώσει άμεσα αποτελέσματα ορατά είναι να βλέπουμε ποιε πρωτοβουλίε αναλαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, εθνικό επίπεδο. Να δούμε τι έχει αποτέλεσμα και θα είμαστε σε θέση να δούμε τα αποτελέσματα των διαφόρων μέτρων μόνο σε μερικά χρόνια. Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι για μια κατηγορία, τους βετεράνους, για αυτή την κατηγορία δεν είναι δυνατότητα να, δεν υπάρχει δυνατότητα να δείξουμε ίκτο. Ερχόμαστε τώρα στην ερώτηση του Τσέχου Ευρωβουλευτή. Δεν επιτιθέμεθα κατά ιδεών. Μιλάμε για ποινικά δικήματα. Εγκληματίες που χρησιμοποιούν τη θρησκεία για να διαπράξουν εγκλήματα με τρομοκρατική πρόθεση. Αυτό αντιμετωπίζουμε στις περιπτώσεις των επιθέσεων στο Παρίσι και των, στο, στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Άρα χρειάζεται συνέστημα ευθύνης και συνειδητοποίηση ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Γι' αυτό γίνονται συνεδρία του δικτύου. Και εδώ έρχομαι στην ερώτηση της κυρία Κέρκοφ όχι μόνο θέλουμε κοινή προσέγγιση και να είναι αυτό αυτός σκοπός, θα πρέπει εμείς όμως να κάνουμε τη δουλειά μας. Γι' αυτό θέλουμε το συντονισμό. Παράδειγμα, στις επιθέσεις των Παρισίων και στο μετέπειτα διάστημα χρειαστήκαμε από τις 12 Νοεμβρίου, στις 12 Νοεμβρίου δύο ώρες για να έρθουμε σε επαφή με όλους τους NCT. Να τους ζητήσουμε να τελούν εν αναμονή. Ούτως σε πραγματικό χρόνο να μπορούσουμε να κάνουμε τα δέοντα για δικαστική συνεργασία. Περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό έχουμε το δίκτυο. Και ποια είναι τα καλά μαντάτα. Στις 22 Μαρτίου με ενημέρωσαν σε πραγματικό χρόνο από τις βελικές αρχές και αμέσως σε μισή ώρα ήταν σε αναμονή όλο το δίκτυο. Και ήρθαμε σε επαφή με τους αρμόδιους. Αυτό πρέπει να επιδιώκουμε είναι ένα κομμάτι της καταπολεμήσεως της τρομοκρατίας. Θέλουμε το NCIS να λειτουργεί στο σύστημα εθνικού συντονισμού. Κύριε Βος, ασχολείστε με τον κανονισμό για το Eurojust. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για θέμα τρομοκρατίας. Το NCS θα συμμαζεύει τους NCTs γρήγορα. Το Eurojust ενεπλάκει στις επιθέσεις των Παρισίων και των Βρυξελών. Τι κάναμε. Εξασφαλίσαμε ταχεία δικαστική απάντηση όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία που πετύχει σε πραγματικό χρόνο. Συντονίσαμε τους αρμοδίους και εξασφαλίζαμε σωστά απαντώντας στις ανησυχίες του κ. Βανκερχόφ. Ε, σε κοινέ ερευνητικές ομάδες, να τις μαζεύουμε γρήγορα και είδαμε αύξηση των αριθμών αυτών των ομάδων με τις επιθέσεις των Παρισίων. Αυτό είναι, αυτή είναι η ρόλη ζωές μας. Είναι η ταχεία της αμοιβές δικαστικής αρρωγής. Τι προσφέρουμε. Πρακτική υποστήριξη, δικαστική υποστήριξη, νομική τι αυτή, οικονομική τι αυτή. Διότι έχουμε τεχνογνωσία στο Eurojust. Αξιολογούμε πόσο αποτελεσματικοί είμαστε. Σταθερά, κάθε χρόνο. Συνεδρίαση του δικτύου με εκπροσώπους αστυνομία και του δικαστικού κλάδου και των κρατών, όλων των κρατών μέλων. Αυτό κάνουμε συνεχώς. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση τη κυρία Είναι πολύ σημαντική η οδηγία. Γιατί? Διότι εμείς αυτό που κάνουμε είναι να στοχεύουμε όχι μονάχα σε ενό είδου τρομοκρατία. Και αυτό είναι το καθήκον μας, γιατί βρισκόμαστε μέσα σε πλαίσιο κράτους συνταγματικού ε, ε, δικαίου. Υπάρχει το δικαίωμα να μετακινείται κανεί, να εκφράζει την άποψή του. Εμεί όμω ω εισαγγελεί έχουμε μία υποχρέωση. Να προστατεύσουμε το δικαίωμα στη ζωή. Εάν παραβιαστεί αυτό το όριο, τότε καλούμαστε να δράσουμε και να αντιδράσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό ε, από την δικαστική άποψη και προληπτικά. Γι' αυτό χρηματοδότηση γι' αυτό ε, η αντιμετώπιση των ταξιδιών που έχουν τρομοκρατικό σκοπό. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Αν πας στην Συρία όχι για διασκέδαση, όχι για ψυχή, αλλά για να ανακατευτεί σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Στρατολόγηση, ε, συστράτευση, ε, προσφορά έμπνευση σε άλλους, ε, διεξαγωγή πολέμου, αποκεφαλισμοί, ομοιρίες δημοσιογράφων μιλούμε για δημοσιογράφους οι οποίοι συλλαμβάνονται όμοιροι στη Συρία. Το άλλο μεγάλο θέμα εδώ είναι πώς βρίσκεις αποδείξεις σε αυτές τις χώρες. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Και γι' αυτό αναζητούμε τρόπους να ενισχύσουμε τους τρόπους με τους οποίες μη ευρωπαϊκές χώρες, ε, χώρες δηλαδή ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν στον τομέα αυτό, όπως χώρες της Εγγύης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, του, των, ε, ε, των Βαλκανίων. Πέρσι, στην τακτική συνάντηση με τους εισαγγελείς και συζητήσαμε με τους 28 αρμοδίους, βάλαμε μέσα την Ορβηγία τις ΗΠΑ και την Ελβετία. Επίσης όμως την Τουρκία, τα Δυτικά Βαλκάνια και τους Τινήσιου. Γιατί του Τινήσιου είμαστε ήδη αναμειγμένοι στην προσπάθεια διαλεύκανσης των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Τινησία που προκάλεσαν σημαντικούς αριθμούς θυμάτων. Άνθρωποι οι οποίοι μεταβαίνουν στην Τινησία για να ξεκουραστούν στην παραλία είναι οι άνθρωποι που μας απασχολούν. Είναι τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Αυτά δεν πάντα κάνει μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να συνεργαστεί με επαγγελματίες επιτόπου και χρειάζεται να τα κάνει όλα αυτά μέσα στα πλαίσια του κράτους δικαίου. Τώρα μετακινείται, τώρα, μετακινείται οι, ε, ε, μετακινούνται οι τρομοκράτες από την Τιτσία στη Λιβύη. Είναι εύκολα τα πράγματα αυτά, όχι δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Χρειαζόμαστε χρόνο. Αλλά βεβαίως πάντοτε με μια αίσθηση κατεπίγοντος. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας λοιπόν. Και σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, βλέπουμε πολλούς ανηλίκους, η προστασία των παιδιών είναι πολύ σημαντική υπόθεση για μα. βλέπουμε σε κάποιες χώρες να είναι δυνατό να γίνει δίωξη, να είναι δυνατό να καταδικαστούν τα πρόσωπα αυτά και εν απουσία τους, ερήμην. διότι καμιά φορά χάνουν τα τους και μετά, α, εντελώς τυχαίως επανέρχονται σε κάποια τρομοκρατική επίθεση. Δεν είναι στη βάση μόνο πληροφοριών τα όσα κάνουμε. Είναι και στη βάση ενός πραγματικά, μιας πραγματικά λεπτομερούς δικανικής εργασίας. Και πάντα με νόμιμο τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται οι δικαστικές αρχές με τις αστυνομικές αρχές. Όπως είπα, σε, μέσα σε νομικά πλαίσια. Πράγματι, για να εστιάσουμε και θυμίζω εδώ το άρθρο 13 της απόφασης της Eurojust να είμαστε τακτικά ενημερωμένοι και για άλλες μορφές εγκλημάτων. Κύριε Βόση, έχετε δίκιο. Είδαμε συνεργασία, διασύνδεση μεταξύ τρομοκρατών και εγκληματιών του κοινού ποινικού δικαίου είτε πρόκειται για ε, δουλεμπόριο, διακίνηση προσώπων, είτε πρόκειται για χρηματοδότηση και μιλούμε και για επαναστατικούς φόρους, για οργανωμένο έγκλημα και για ε, δραστηριότητες ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεπτόμαστε και να αρχίσουμε να εργαζόμαστε και εκτός πλαισίων και όχι πάντα μέσα στα πλαίσια. Διότι υπάρχουν και αυτοί που ε, βγαίνουν εκτός πλαισίου και δεν είναι όλοι μόνο ιδεολόγοι τρομοκράτες. Υπάρχουν και οι κοινοί ποινικοί οι οποίοι συνεργάζονται μαζί τους. Επανέρχομαι στην ανησυχία του κ. Κάρκοπ. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των χωρών μελών και εκεί ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, αλλά να εξασφαλιστεί ότι η Eurojust μπορεί να κάνει και διασταύρωση των πληροφοριών. Το κάνουμε αυτό σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, που είναι στην ουσία ο βασικός μας εταίρος και το γεγονός ότι έχουν φτιάξει το Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με την Ευρωπόλ. Και αυτό κάνουμε άλλωστε με την ε, συνθήκη. Ε, έχουμε έναν ε, απόλυτα εξειδικευμένο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος διασφαλίζει τη συνεργασία με την Ευρωπόλ. Και την δικαστική συνέχεια που δίνεται στις προφορίες που συλλέγει η Ευρωπόλ και μέσω των άλλων κέντρων συντονισμού. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Γκίνσπερκ για τις ε, ερωτήσεις της. Α, με συγχωρείτε. Καλά, τότε λοιπόν θα ολοκληρώσω και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα αφού μου το ζητεί ο πρόεδρος σας. Πράγματι, η δικτύωση των τρομοκρατών πρέπει να βρει απέναντί της τη δικτύωση δική μας. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για θέματα τρομοκρατίας και αντιτρομοκρατίας που δίνει αρχίσει και δείχνει τα δόντια της με τις καταδίκες αρχίζουμε και πετυχαίνουμε καταδίκες αναλύουμε τις καταδίκες μέσα από τα δίκτυά μας με τη λεπτομερή ανάλυση εμβληματικών καταδικών θα ήθελα να σας δείξω και βελγικές καταδίκες που αποτέλεσαν πηγή έμπνευση για πρόσφατες ισπανικές καταδίκες. Και τα αναλύουμε όπως είπα αυτά και τα συζητούμε στις συναντήσεις μας. Αυτό κάνουμε στην ουσία. Και αυτό κάναμε και σε πτυχές ε, εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Έχουμε ένα αριθμό φακέλων που μας έρχονται μέσα στα πλαίσια της ατζέντα της ασφάλειας για θέματα τρομοκρατίας κτλ. όπου η Eurojust παίζει ένα σημαντικό, αν και περίπλοκο ρόλο. Θα σας ζητήσουμε λοιπόν, όταν συζητήσουμε κάποια από τα θέματα αυτά σε διάφορες ακροάσεις, ε, να συνεργαστείτε μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, καθώς και για την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε και βεβαίως είστε πάντοτε σε επαφή με τα πιο πρόσφατα γεγονότα. Σας ευχόμαστε και καλή τύχη και σας ευχαριστώ και πάλι αγαπητή Μισελ για την έλευσή σας και την παρουσίαση στην οποία προέβητε. Σας ευχαριστώ κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Στις 3 συνεχίζει τη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ.